Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Sitzung. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλημέρα σας. Με την Tagesordnung eine... Κρίση της διάταξης. Ε, προτείνουμε μια αλλαγή που είναι απαραίτητη. Το αεροπλάνο από την Κοπεχάγη έχει καθυστέρηση μία ώρα. Οπότε η κυρία Ζακλίν Μακλέιτ θα φτάσει κατά τις 4 και όχι κατά τις 3. Τι κρίμα. Έχουμε όμως και άλλα θέματα στην ημέρα στη διάταξη και μπορούμε να το μεταθέσουμε. Δεν θα μας απο... Ε, κλείσει ή θα μας αποτρέψει από τις εργασίες μας αυτό. Και αφού είναι εδώ οι συνάδελφοι των επομένων θεμάτων, μπορούμε να αλλάξουμε το 4 και το 5 να προταχθεί και μετά να συνεχίσουμε με το 3 όταν φτάσει με το καλό η κυρία Μακλέιτ. Φαντάζομαι ότι δέχεστε την ημέρα σε διαταξή με τις τροποποίησεις αυτές. Ανακοινώσει του Προέδρου. Να σας πω για το εργαστήρι, workshop. Την Τετάρτη, για το 2050, ε, για τις χαμηλές εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, ο Κρίς Ντέβις προεδρεύσει. Παρακαλώ να είναι αρκετά μέλη της Επιτροπής Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει. Η Γαλλική Συνέλευση στο Παρίσι αποφάσισε να απαγορεύσει τη βυσφενόλη α για ε, προϊόντα που προορίζονται για βρέφη. Νομίζω μετά τη Δανία Γαλλία είναι η δεύτερη χώρα που το απαγορεύει και είναι ένα πάγιο μέλημα της Επιτροπής μας να απαγορεύεται η χρήση αυτής της ουσίας στα βρεφικά είδη. Λοιπόν, φτάνουμε ήδη στο σημείο 4, αφού μεταθέσαμε το 3, που είναι προφορική ερώτηση. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κυρίας Λεπάς και του κυρίου Γκερμπράντη για τις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για λιπογόνες και μη βιώσιμες πρακτικές. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση απόπειρα αλλά δεν μπήκε τελικά στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας γιατί έτσι εδέησε η διάσκεψη των Προέδρων, παρήλθε η προθεσμία μετά από τρει μήνε και αποφάσισαν οι συντονιστέ να αρχίσουν από την αρχή την προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω, Κορίν ή ο Γερμπράντη, κάποιο από του δύο να παρουσιάσει την ερώτηση και μετά να ψηφίσουμε και τυπικά ότι θα το επαναφέρουμε το θέμα προσυζήτηση είναι ερώτηση. Η κυρία Λεπάζ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντω είναι η δεύτερη απόπειρα, όπως θυμήσατε, που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περί τίνος πρόκειται, απλούστατα. Και για να είμαστε τυπικοί και ε, πειθαρχημένοι από πλευρά του προπολογισμού μας που ενδιαφέρει όλου μα, αλλά και να είναι αποτελεσματική η δημόσια δαπάνη, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται με τι επιδοτήσει, που στην πραγματικότητα βοηθούν στη ρήπανση. Δηλαδή από τη μια πληρώνουμε για να καθαρίζουμε και από την άλλη πληρώνουμε για να ρηπαίνουμε. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μια συνολική θεώρηση, να δούμε τι επιδοτήσεις πηγαίνουν στη ρήπανση για να μπορέσουμε λίγο να τις περιορίσουμε ω προ το ποσό και να μην ε, πηγαίνουν τα κοινοτικά κονδύλια εκεί για να πιάνουν τόπο αλλού. Το Συμβούλιο κατά τα άλλα πρέπει να σα πω έχει πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος γιατί είναι και στη δική του ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι είναι σημαντικό εμεί, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εργαστούμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει σε πέρα σε αυτή την προσπάθεια, να μας καταθέσει μια αξιολόγηση των επιδοτήσεων που είναι ρηπογόνες και να καταργηθούν εκείνες που οφείλουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσει τα χρήματα ο κλάδος της οικονομίας. Θα πηγαίνουν στον ίδιο κλάδο, αλλά για άλλη χρήση. Όχι για τη ρηπογόνα. Αυτό είναι νομίζω το γενικό συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ, Κόγιν Λεπάζ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Γκερμπράντι, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Yes, thank you, Chairman. I don't have... Ναι, ευχαριστώ, πρόεδρε. Στα αγγλικά δεν έχω να προσθέσω πολλά. Μόνο ότι σε αυτού του καιρού τη λιτότητα θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα να μην ε, σπαταλώνται αυτά τα κονδύλια με τον τρόπο που γίνεται σήμερα με τις επιδοτήσεις που πηγαίνουν για ρηπογόνα πράγματα. Τώρα πλέουμε δύο φορές. Δίνουμε επιδοτήσεις για να ρηπαίνουν και μετά δίνουμε επιδοτήσεις για να καθαρίζουμε ε, και να επανορθώνουμε τις ζημίες. Ε, η πολιτική λοιπόν ανάγκη και το επίγον ε, είναι δεδομένο. Θα πρέπει να επαναλάβουμε αυτή την προφορική ερώτηση και στη συνέχεια ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη διάσκεψη των Προέδρων για να μπει και το θέμα τη μέση διάταξη ολομέλης. Ναι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη αυτή και έγκυρη ερώτηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ενεχομένους που παίρνουν ε, επιδοτήσεις για ρηπογόνες πρακτικές. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν αυτής της προφορικής ερώτησης. Thank you. Who is against? Κατά. Αποχές σαφής πλειοψηφία υπέρ. Uh, Άρα θα μπει στην Ολομέλεια. Ωραία. Θα το υποβάλουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ και πάμε στο σημείο 5. Η Άννα Ρόσπαχ ε, έχει έρθει. Οπότε μπορούμε πιο εύκολα να ασχοληθούμε με το θέμα. Πώ θα αποφευθεί η σπατάλη τροφίμων, στρατηγικέ για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα τη τροφική αλυσίδα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό το θέμα για την αποτρασματική χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και την επισητιστική ασφάλεια παγκοσμίω, αν μη τι άλλο στην Ευρώπη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο μέσω στην εισηγητρή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Έχω Διάβασα την ε, έκθεση της συναδέλφου Καρόνα, Κούρονα, η οποία και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ασφαλώς και διδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, μέχρι 50% των τροφίμων στην Ευρώπη ουσιαστικά για διάφορους λόγους ε, πετιούνται. Και αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά αποτελεί και κάτι αντιδιοντολογικό και από πλευρά ενεργειακή επίσης δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πετάμε τρόφιμα. Τα προβλήματα λοιπόν παρατηρούνται σε, διάφορες, σε διάφορα επίπεδα και σε ό,τι αφορά και την παραγωγή των τροφίμων, αλλά και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές τις μεγάλες κουζίνες, τις καντίνες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Βόρεια Αμερική. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι σπατάλες γίνονται πιο πολύ κατά την παραγωγή και κατά τη μεταφορά κυρία Καρόνα αναφέρει ότι είναι περιορισμένε οι δυνατότητέ μα σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτό. Εγώ θεωρώ όμω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιούμε καλύτερα τα τρόφιμα που έχουμε στη διάθεσή μα. Η κατανάλωση τροφίμων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο παραγωγής. Άρα οι υπερητέ μεταφορέ, ε, όπορο λαχανικών και κρέατος θα πρέπει να αποφεύγονται όπου αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, 2,3 τόνοι ψάρια πετάμε κάθε χρόνο. Αυτό αποτελεί μεγάλο ποσοστό των συνολικών ε, του συνολικού ε, ψαριού που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά οφείλονται σε σφάλματα που γίνονται μεταξύ 20 και 30% της συνολικής παραγωγής όπορα λαχανικών πετιούνται για αισθητικού λόγους. Επειδή δεν ανταποκρίνονται στι αισθητικέ μας προδιαγραφέ σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, και τα αγκουράκια. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να ενημερώνουν τα καταναλωτή. Από τον βρεφονιπιακό σταθμό θα πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά ότι τα τρόφιμα αποτελούν ένα πόρο τον οποίο θα πρέπει να εκτιμούμε, να επανέλθουμε σε έναν τρόπο σκέψης και ενέργειας όπως οι νοικοκυρές, προκειμένου να μην καταλήγουν όλα στα σκουπίδια. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να διαβάσετε αυτά που έγραψα. Έγιναν και κάποιες ε, τροπολογίες από τους συναδέλφους και η προθεσμία είναι την Τετάρτη στις 12. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Όχι μόνο ρηπαίνουμε τα ύδατα, αλλά πετάμε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πιο υπεύθυνο τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε, Άννα Ρόσπαχ, για το σχέδιο γνωμοδότησης, για την ε, έκθεση της ε, Επιτροπής Γεωργίας και ανάπτυξη της πέτρου. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Όντω, το 4 αναφέρεται ότι κάποιες απαιτήσει ποιότητα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι απαιτήσει ε, που οδηγούν τελικά σε απόρριψη πολλών τροφίμων. σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει, δηλαδή της αγοράς, που ίσως να μην έχουν να κάνουν απαραίτητα με τα κριτήρια ε, χρησιμοποίησης ή μη των τροφίμων. Γίνεται στην Γερμανία μια συζήτηση για την ημερομηνία ανάλωση. Έχει γίνει και μεγάλη τηλεοπτική συζήτηση για το κατά πόσον είναι παραπλανητική αυτή η ημερομηνία γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και ίσως θα ήθελε να τοποθετηθεί και από αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον υπάρχουν κάποιοι νόμοι ή κατά πόσον ακολουθούνται πρακτικές της αγοράς και πώς θα μπορούσαμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο, ο Ρίχαρτ Ζέιμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να, να πω ποια είναι η θέση της Ρενάτε Ζόμερ αυτή η εκπροσωπώ γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Ευχαριστώ την Άννα Ρόσμπαχ για την ε, κατάρτιση της γνωμοδέτησης. Διαβάζοντας την γνωμοδότηση αυτή πραγματικά ντρέπομαι γιατί βλέπουμε πόσο τρόφιμα καθημερινά πετάει ο καθένας μας στατιστικά. Μιλάμε για την ε, βιομηχανική μας κοινωνία για κάτι πραγματικά επέσχυντο. Έχουμε διάφορους μηχανισμούς για τα σημαντικά όμως αυτά προβλήματα δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν έχουν βρεθεί οι σωστές λύσεις, ιδιαίτερα κοιτώντα ε, και την αυξητική τάση από τη δεκαετία του 70. Πραγματικά αυτά προκαλούν ε, ένα δυσάρεστο συνέστημα, όπως ξέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών, το πρόβλημα είναι στην κατανάλωση και στην διανομή. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει εκεί να επικεντρωθούν οι προσπάθειές μας. Και σωστά αναφέρει η κυρία Ρόσπαχ τι μπορούμε να κάνουμε. Ότι καταρχάς θα πρέπει να γίνει ένα awareness raising, να αναπτύξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και σε ό,τι αφορά αυτή την ημερομηνία ανάλωση. Σε πολλές περιπτώσεις είναι παραπλανητική. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με τρόφιμα όπως τα λαχανικά και τα φρούτα. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν θα ήθελα να εκφράσω την απόψή μου για τέτοια φαινόμενα, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να πείσουμε τον καταναλωτή να αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα αυτά τα τρόφιμα. 13%. Α, συγγνώμη, 30% το 1 τρίτο των συσκευασμένων προϊόντων το πετάμε κατευθείαν χωρίς να το βγάλουμε καν από τη συσκευασία του. Είναι απίστευτο. Και το τι σημαίνει αυτό φυσικά και για το ενεργειακό κόστο. Ο κόσμος φυσικά έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει τι καθημερινέ του ανάγκε και νομίζω ότι καλό θα ήταν η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει πιο έντονα και εντατικά το θέμα αυτό και οι συνάδελφοι να σκεφτούν τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχά, για να γίνει αυτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κατά δεύτερον, για να ερευνήσουμε πώ ε, στο εμπόριο μπορούμε να ακολουθήσουμε προσεγγίσει ε, για να αξιοποιούνται καλύτερα τα τρόφιμα, πώ μπορούν τα τρόφιμα αυτά να καταλήγουν σε ομάδες ε, του κόσμου που τα χρειάζονται. Το δεύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αναπτυξόμενες ε, χώρες και τις χώρες ανάπτυξης που έχουν ε, προβλήματα αντίστοιχα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μέσω μεταφοράς ε, τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, την ψήξη στην μεταφορά, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος. Στο μέλλον, ο Παγκόσμιο πληθυσμό θα φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια. Άρα το θέμα αυτό θα καταστεί ακόμα πιο ε, σημαντικό και κατεπήγον. Και νομίζω ότι εμεί ω Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει σίγουρα να συμμετάσχουμε. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Ρόσμπακ, αλλά παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πιο έντονη δράση στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, Λίντα Μακέβαν. Είμαι, ο σκιώδης μα δεν είναι εδώ ούτε αυτός, οπότε θα κάνω κάποια σχόλια. Ευχαριστώ την Άννα για την έκθεσή της. Είναι σημαντικό το θέμα. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, όπως στην Γερμανία, συζητείται πολύ το χρέος και η κυβέρνηση θα αλλάξει το νόμο. Θα απαγορεύσει, α, της ημερομηνία μόνο το πρόβλημα. Θα λένε χρήση μέχρι την τάδε ημερομηνία και όχι ημερομηνία πώληση, ποια είναι τελική ημερομηνία πώληση, ε, τελική ημερομηνία χρήση και για κροσέρβες και λοιπά συσκευασμένα θα λένε ότι είναι καλύτερα πριν, να καταναλωθούν πριν από την ημερομηνία. Αυτό δεν έχει επιστημονική βάση. Και είναι κάτι που δεν θα πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι καλό το προϊόν ακόμα και όταν η ημερομηνία που αναφέρει ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση μετά την ημερομηνία δεν ισχύει. Και μπερδεύουν τους ε, πελάτες. Μετά τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ πώς πολλούν οι λιανοπολιτές. Σε πολύ μικρό σούπερ μάρκετ στην περιοχή μου το συζητούσαμε. Για τον Αρακά ήθελα ένα πακέτο μόνο. Και μου λένε όχι θα αγοράσετε δύο στην τιμή του ενός και λέω όχι δεν θέλω, θέλω να έχω ένα πακέτο, όχι να πάρετε το άλλο, χρειάζεστε δύο στην τιμή του ενός. Αυτή είναι κοινή πρακτική. Προσφορές δύο στην τιμή του ενός. και η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν παίρνουν το κέρδος οι παραγωγοί, αλλά το κέρδος το παίρνουν οι λιανοπολιτές. Πιέζονται να παράγουν τη διπλάσια ποσότητα για τις προσφορές 2 για 1, αλλά δεν καρπούνται το κέρδος. Θα ακούσατε πολλές διαμαρτυρίες όταν αφορά γι' αυτό, οι ηλικιωμένους, αυτούς που μένουν μόνοι, που είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν μεγάλα πακέτα ε, με λαχανικά και θέλουν λίγα. Θέλω να είναι πολύ δύσκολο σε μεγάλο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν ένα-δύο καρότα, ένα-δύο κρεμμύδια κλπ. Υπάρχουν και οργανώσεις που διανέμουν τρόφιμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία που αναφέρει στη συσκευασία ότι είναι καλύτερο να καταναλωθούν μέχρι τότε. Και είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δει πώς μπορούν να χρηματοδοτούνται αυτές οι οργανώσεις για να μην πετιέται το φαγητό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται μιλάμε για σπατάλι που, ε, μιλάμε για τα τρόφιμα που δεν μπορούν να φαγωθούν μετά καθόλου, να καταναλωθούν. Ε, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιομάζα. Οι κυβερνήσεις πλησιάζουν το θέμα περίεργα. Δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα απόβλητα για παραγωγή βιομάζας. Εισάγουν υλικό το χάρη παρθένα δάση αν δεν χρησιμοποιήσουν βιομάζα θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα της κοινωνίας για αυτό το σκοπό. Το εξετάζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποτίθεται θα μας δώσει κάποια βιώσιμα κριτήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλά τέτοια τρόφιμα που είναι για τα σκουπίδια μπορούν να χρησιμοποιούνται για βιομάζα. Και να δούμε και τι γίνεται στο κτίριο του Κοινοβουλίου με τα απόβλητα. Πας πολλές φορές σε μια δεξίωση και μένει πολύ φαγητό. Πού πάει θα έπρεπε να στείλουμε στις, ε, στην, ε, στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μάθουμε πού πάνε αυτά τα τρόφιμα και θα ξέρουμε πού καταλήγουν αυτά τα τρόφιμα. Στο Στρασβούργο ξεχωρίζουμε, διαχωρίζουμε και βάζουμε σε τρει διαφορετικούς κάδους τα σκουπίδια μας και μετά έρχονται οι καθαρίσεις και τα βάζουν όλα σε έναν κάδο και φεύγουν. Πρέπει να γράψουμε λοιπόν στι αρχέ του Κοινοβουλίου και να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει με τα τρόφιμα εδώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Ε, στη χωματερή θα πηγαίνει ή στην αποτέφρωση, δεν ξέρω. Συχνά ε, γίνονται συζητήσεις κατά τη διάρκεια του γεύματος με όλα αυτά τα ωραία σάντουιτς που μετά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Παίρνουν σε μια μεγάλη σακούλα και από εδώ πάνε κι άλλοι. ούτε τα ε, ανακυκλώνουν ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, κάρτη καλλιωτά. Ε, Ευχαριστώ. Γιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Άννα Ρόσμπαχ για την έκθεσή της. Την γνωμοδότηση καλύτερα. Και ε, συμφωνώ και με τους προαλαλήσαντες που είπαν ότι η απόρριψη των τροφίμων είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κρίμα. Στον τελικό καταναλωτή, αν δείτε τι γίνεται, χρειάζεται τεράστια αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να δούμε πώς σκέφτεται ο κόσμος και πώς ε, πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε ε, στο μέλλον. Βραχυπρόθεσμα όμως αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε κάποιες λύσεις ε, όπου είναι σχετικά απλό να υπάρξουν βελτιώσεις. Παράδειγμα, στην αλυσίδα παραγωγής, στη φάση ε, της ε, ε, τυποποίησης και διανομής υπάρχει πολύ μεγάλη σπατάλη τροφίμων. Καταλαβαίνω για λόγους αισθητικούς ή οικονομίας χρημάτων ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική για τα απορρίμματα τροφίμων και τα βιολογικά και να ξέρουμε ότι η καλύτερη αντιμετώπιση των απορριμμάτων είναι η πρόληψη. Και για τα τρόφιμα ισχύει αυτό και ε, έχει να κάνει με ε, την παραγωγή αρίων ε, θερμοκηπίου κατά όλη την αλυσίδα της παραγωγής, με την κατανάλωση ύδατος και άλλα τέτοια προβλήματα που πρέπει να αποφύγουμε και να προλάβουμε. Εκτός αυτού, είμαι υπέρ της δωρεάν διανομής τροφίμων Βέβαια, δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να ε, το έχουν αυτό ως αντανακλαστικό κοινωνικής πρόνοιας, ότι εντάξει άποροι θα τους με τα τρόφιμα που έτσι κι είναι για πέταμα. Σε καμία περίπτωση. Και... Επίσης, ε, γίνεται μεγάλη κερδοσκοπία ε, στις καλλιεργήσιμες γέες, τεχνητά υψηλές οι τιμές των τροφίμων και πολλές φορές για τους καταναλωτές είναι πολύ πιο φθηνό να πετούν τρόφιμα που είναι καλά προς, προς κατανάλωση. Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια για τις ποσοστώσεις του γάλακτος τι έγινε. Πώς πετούσαν ε, το γάλα στο δρόμο οι κτηνοτρόφοι. Και εντάξει μπορεί κανείς τότε να τους καταλάβαινε αλλά 995 εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη σήμερα υποσυντίζονται. Και είναι σκάνδαλο που υπάρχουν ακόμα ευρωπαϊκοί κανόνες και επιτρέπουν κάτι τέτοιο την απόρριψη έτσι τροφίμων και να είναι πιο οικονομικό και πιο κερδοφόρο το να ε, καλλιεργείς για τη χωματερή παρά να ε, διαθέτεις τα τρόφιμα εκεί που πρέπει. Χρειάζεται καλύτερη εστίαση και περιορισμός αυτού του φαινομένου Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρος στα Ολλανδικά. Ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Άννα Ρόσμπαχ για το κείμενό της θα σας ενοχλήσω. Με ένα κολπάκι που χρησιμοποιούσαν οι γονεί μου όταν θέλαν να δουν ένα φρούτο ήταν ακόμα ε, θα μπορούσε να φαγωθεί, το δίναν στη γάτα ένα κομμάτι και αν το ήθελε η γάτα ήταν ασφαλές το φαγητό, αν δεν το ήθελε δεν ήταν ασφαλές διότι τα ζώα ξέρουν. Δεν έχουν όλοι γάτο όμως. Ίσως ε, μπορούμε με νέα τεχνολογία να βρούμε έναν τρόπο. Ίσως έτσι θα μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια γάτα του 21ου αιώνα. Τι έχω υπόψη μου. Νανοτεχνολογία. Υπάρχουν τρόποι ούτως ώστε στην συσκευασία να μπει κάτι και να μην αποφασίζει η αναγραφόμενη ημερομηνία θα πετάξει το φαγητό είτε όχι, αλλά η συσκευασία θα δείχνει κατά πόσο είναι ασφαλές προς κατανάλωση. Ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιομηχανία το εξετάζει το θέμα. Αυτοί εξετάζουν το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία και ούτω τρόπος να βοηθηθούμε ούτως ώστε να μειωθεί αυτή η σπατάλη των τροφίμων. Ευχαριστώ. Η δοκιμή της γάτας είναι διεθνής, το κάναμε και εμείς στη Γερμανία. Πού να δείτε η γάτα μας, εμάς δοκίμαζε αν ήταν το γάλα εντάξει ακόμα καλό και άλλα πράγματα, όχι μόνο στην Ολλανδία έτσι. Ο Ρώση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Άννα Ροσμπά και την έξοχη δουλειά που έκανε. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα, όπω και σε άλλε χώρε ενδεχομένω, μπορεί να είναι και η αλλά συγκεκριμένα στην Ευρώπη υπάρχει μια υπερβολή σπατάλη ε, φαγητού. Πολύ συχνά πολλούνται πολύ μεγάλες δόσεις και πρέπει να προσέχουμε ζητάμε και πολύ λίγα. Διότι υπάρχει και αντίστροφη όψη του νομίσματος. Πολύ μικρές ποσότητες, πολύ συχνά μπαίνουν μέσα σε πολυστερίνη ή σε νάιλον σε συσκευασία και μετά ε, θα πρέπει αυτά να πάνε στα απόβλητα. Και καμιά φορά στον καταναλωτή κοστίζει περισσότερο αυτό. Να πληρώνει μια τέτοια συσκευασία που πετά παρά να έπαιρνε μια ποσότητα ε, προϊόντος μεγαλύτερη. Και ε, ίσως και γι' αυτό όμως τελικά να αγοράζονται πολλά τρόφιμα. Από τα μπουφέ του Κοινοβουλίου δεν νομίζω να πετιούνται πολλά, Πρόεδρε. Πέρα που είμαστε πολύ, ε, ε, έχουν πολύ λίγα τρόφιμα και κοστίζουν και πολύ εξάλλου. Πιστεύετε ότι αν θέλει να, να φέρει κανείς για να, τις, να φέρει από την περιοχή του τα μπουκάλια ε, για να τα ανοίξει εδώ πρέπει να πληρώσει 4 ευρώ ε, τέλος ε, ανοίγματος αν θέλετε εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι φέρνουν πολλά και πετιούνται πολλά. Πολύ συχνά μεγάλες αλυσίδες διανομής ε, πετάνε πολλά, όπως η McDonald's. Παράγει πολύ καλά προϊόντα και εγώ πάω συχνά στο McDonald's, αλλά το λένε και οι ίδιοι δυστυχώς, ότι έχουν ένα πολύ αυστηρό κανονισμό πρέπει να σέβονται. Τα ψωμάκια πετάγονται μετά από 10 λεπτά από την παραγωγή. Μπορούν να μείνουν αναμονή τα έτοιμα ψωμάκια μόνο 10 λεπτά σπατάλει τεράστια προφανώς τροφίμων. Ε, είναι αδίκημα. Σκεφτείτε οι άλλοι δεν έχουν τρόφιμα και εμείς σπαταλάμε τρόφιμα που είναι καλά και πάρα πολύ καλά που θα μπορούσαν να φαγωθούν. Αυτό πονάει, κάνει κακό. Άρα θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βρούμε, και αυτό ζητά από την Άννα Ρούσμπαχ, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην Ιταλία υπάρχει τράπεζα τροφίμων. Νομίζω ότι υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες που μαζεύουν τα φαγητά, τα τρόφιμα, ασχολούνται αυτοί οι φορείς, βλέπουν αν μπορεί να φαγωθεί το τρόφιμο, εάν έχει λήξει η προθεσμία κατανάλωση, η ημερομηνία κατανάλωσης, ή με επαγγελματίε να παληθεύουν και κάνουν αναδιαμονή, α, διανομή δωρεάν σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Διότι κάθε μέρα πετάμε τόνους καλού φαγητού. Αν καταφέρουμε λοιπόν να αφήσουμε στην κυκλοφορία και δίνοντας αυτά τα φαγητά σε αυτούς που χρειάζονται τα τρόφιμα κάνουμε έξοχη δουλειά για εκείνου που έχουν ανάγκη και ζητώ από την Άννα αν θα ήθελε στην έκθεσή της να, κάνει και αυτή την πρόταση για να βοηθήσουμε αυτούς τους φορείς, αυτές τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη συλλογή αυτών των τροφίμων και να αποφύγουμε τις πατάλες. Όχι μόνο αυτό, θα μπορούσαμε Πρόεδρε, μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς, να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε μια εξοικονόμηση όσον αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Διότι είναι, μια άχρηστη σπατάλη από την άλλη πλευρά, αλλά να πετάγονται και στα σκουπίδια είναι ε, και κακό και για τι ε, χωματέρε. διπλό κακό. Γιατί μπορούσαμε να δώσουμε και δωρεάν φαγητό σε αυτού που έχουν ανάγκη. Ο ευχαριστώ. Ναι, όλοι οι συνάδελφοι έχουν δίκιο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γάτα. Αυτό που ε, προκαλεί έκπληξη είναι ότι έχει επισέλθει αυτή η συνήθεια, γιατί ε, εμεί είχαμε τη γάτα. Τα παιδιά μου, τι να σας πω, έχω απετύχει τελείω. Αν τα παιδιά μου ε, πάρουν μαζί στο... Πέραν μαζί στο, στο σχολείο ένα γιαούρτι που είχε, λήξει, είχε περάσει η ημερομηνία του για μία μέρα, ήμουν εγώ ο κακός. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτή την ημερομηνία ανάλωσης. Ποιος την ορίζει, να το δούμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι οι καταναλωτές απέχουν παρασάγκας. Πρόκειται, μάλλον δεν είναι σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές αυτοί που το ορίζουν. Τα καρτέλ μάλλον έχουν συμφέροντα σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών τους ε, για να δημιουργείται η εντύπωση ότι στην αγορά διατίθενται μόνο τα πολύ πολύ φρέσκα προϊόντα Εγώ θεωρώ ότι έχουμε και παράγουμε προϊόντα τα οποία αντέχουν και αποθηκεύονται για μήνες, όπως οι πατάτες, αλλά ένα μόνο μήλο να βρεθεί που να είναι χαλασμένο, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ποιοι ορίζουν λοιπόν τις ημερομηνίε ανάλωσης. Και ύστερα υπάρχει κι άλλο ένα πολύ περίεργο θέμα, ένας περίεργος κλάδος, ο οποίος φροντίζει τα τρόφιμα που βγαίνουν στην αγορά να μην πηγαίνουν στις χωματερές αλλά στις ζωοτροφές. Και αυτή ο κλάδος λοιπόν παίζει ρόλο γιατί φυσικά και τους συμφέρει να επηρεάζουν τις ημερομηνίες ανάλωσης των προϊόντων. για να περνάνε, για παράδειγμα, τα ψωμιά τα οποία ε, αφαιρούνται από τη συσκευασία τους στις ζωοτροφίες, στις ζωοτροφές. Και αυτά λοιπόν μας δυσκολεύουν. Να σας πω ότι δεν έχω ασχοληθεί επαρκώς ακόμα με την ε, γνωμοδότηση αυτή, με την έκθεση αυτή ε, και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, το θέμα της ημερομηνία ανάλωσης. Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την ε, συνήθιση μας, αν θέλετε, την νοοτροπία μας, τις συνήθειές μας, να τρώμε ένα γιαούρτι το οποίο έχει λήξει πριν από μια-δυο μέρες. Ε, κοιτάξτε, αν ήταν κάθε φορά που έτρωγα από το ψυγείο μου στις Βρυξέλλες κάτι που είχε λήξει να αρρωσταίνω, σας το λέω ειλικρινά, δεν θα ήμουν πια υγιής. Ο πρόεδρος, ναι. Πολύ πρόεδρος. Να, προσέχουμε να μας καλεί στο σπίτι σου για φάγη δηλαδή. Ματίας Κότερ. Ματίας Γκρότε, ναι, σας ευχαριστώ. Η Άννα Ρόσμπαχ ε, είπε στην αρχή και μου άρεσε πολύ η αρχική της προσέγγιση, ότι όλα αυτά θα πρέπει να συμβούν στην πρώτη φάση, τα παιδιά. Εκεί θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ε, τα μάθουμε πώς υπεύθυνα θα αντιμετωπίζουν τα τρόφιμα. Και μίλησε για τους νηπιακούς σταθμούς. Ε, η ηλικία αυτή μου ταιριάζει γιατί έχω σήμερα εδώ πέρα ε, καλέσει μια ομάδα προσκεκλημένων που ασχολούνται με τέτοια θέματα και ακούν με μεγάλη προσοχή. Κοιτώντας τα αριθμητικά στοιχεία, 220 εκατομμύρια τόνοι στα βιομηχανικά κράτη ε, πετιούνται. Στη Γερμανία 200, 200 κιλά ανακατακεφαλή και 330 ευρώ αν το μεταφράσουμε σε νόμισμα, σε χρήματα. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κάποια διαδικασία νομοθεσία σε, ό,τι αφορά τα τρόφιμα, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα τροφίμων και την παραγωγή των τροφίμων, σε ό,τι αφορά την ε, απόρριψη τροφίμων και μήπως υπάρχει κάποια τάση η οποία προωθείτε. Αν όχι, θα ζητούσα από την Άννα να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά όλε τι διαδικασίε που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα να εισαχθεί μια τέτοια διαδικασία για το πώ μπορεί να μειωθούν αυτά τα αστρονομικά ποσά, αυτά τα αστρονομικά ποσοστά για να προστατεύσουμε και τον καταναλωτή, γιατί τελικά τα 337 ευρώ που πετιούνται στο σκουπιδοντενεκέ, ανεξάρτητα από σε ποια φάση πετιούνται, πλήττουν και τον καταναλωτή. Κατά δεύτερον υπάρχει μια τεράστια ε, διαφωνία στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές αυτές. Θεωρώ ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα, δηλαδή αυτά που πετιούνται και το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος στην Ευρώπη ο οποίος τα χρειάζεται αυτά τα τρόφιμα για να επιβιώσει, αυτά τα δύο λοιπόν τα άκρα θα πρέπει κάπως να συνενωθούν, να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Η χώρα μου αρνείται να συνεχίσει αυτές τις ε, πληρωμές και λείπει νομική βάση αποφάνθηκε το ΔΕΚ, αλλά θα πρέπει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, να πετάμε λιγότερα και να διαθέτονται σε αυτούς που χρειάζονται. Το είπε και ο συνάδελφος Ρόζη. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα προκειμένου τα τρόφιμα να καταλήγουν σε όσους τα χρειάζονται. Και όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Φλόρεντς, όποιος ε, ίσως ε, κερδοσκοπεί εις βάρος αυτών, να σταματήσει για να μην υπάρχει υπερπαραγωγή, να υπάρχει μια έξυπνη διοχέτευση των τροφίμων αυτών. Προκειμένου να υπάρχει για όλους ε, ε παρκή τρόφιμα και αυτό να καθορίζεται και στη φάση της παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευφύς νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Προφανώς ε, καλωσορίζουμε το νηπιαγωγείο από τη Φρίσλαντ του Ματίας Γκρότα, τους ε, καλεσμένους του και η Κρίστα Κλάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. <clears throat> Ακούγοντας τους συναδέλφους, αναρωτήθηκα σε ποια επιτροπή ήρθα. Γιατί ε, εμείς οι ίδιοι κάνουμε τους κανονισμούς, τις νομοθεσίες, τα πρότυπα, εμείς τα ορίσαμε και τα θελήσαμε. Αυτές οι υψηλέ προδιαγραφές και μέχρι ημερομηνίε ανάλωσης θα πρέπει να είμαστε πολύ αυτοκριτικοί κάθε φορά με τους εαυτούς μας. Το χρησιμοποιεί η ε, βιομηχανία εσκεμένα για να αποποιηθεί και την ευθύνη της. Γιατί αν αγοράσω κάτι και έχει λήξει, Ή μάλλον ε, αν δεν έχει λήξει και έχει χαλάσει το προϊόν, έχω το δικαίωμα να το επιστρέψω και θα πρέπει να το πάρει πίσω ο παραγωγός και ο πολιτής. Θα πρέπει λίγο ε, να τα δούμε αυτά με τους εαυτούς μας. Και όταν ακούω ότι να τα δώσουμε στους απόρους, αλλά δεν τρώνε οι γάτες, για προσοχή λίγο με αυτή τη συζήτηση, να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι και ε, να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, διαθέσιμα για όλους υγιεινά τρόφιμα. Και αρκεί να έχεις λίγο μυαλό και να ξέρεις λίγο από οικιακή οικονομία για να καταλαβαίνεις ε, τι τρώγεται και τι δεν τρώγεται. Και τα υπόλοιπα ότι μπορούν να μαγειρευτούν με άλλο τρόπο, δεν τα πετάμε κατά ανάγκη. Αυτό να ξέρει λίγο από ο νοικοκυριό να σου κόβει λίγο και να έχει και μια αίσθηση για τα πράγματα και μια στοιχειώδη υποστήριξη. Να εκπαιδεύουμε και το πληθυσμό για να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν με τα υπόλοιπα και να μην τα πετάνε. Ε, είναι πολύ μεγάλη η δυνατότητα που έχουμε και το φάσμα εφαρμογής. Και τα τρόφιμα γενικά πρέπει να σας πω είναι πολύ φτηνά. Ε, αγοράζονται σε μεγάλες ποσότητες και αυτό που περισσεύει το πετάμε. Εκεί είναι τα πεταμένα λεφτά και εκεί είναι και πολλές ε, οι δυνατότητες πίεσης. Και ορίζουμε την ποιότητα με τρόπο πάρα πολύ συνειδητό. Ε, εμείς την ορίσαμε αυτή. Και αν πούμε ότι η έσχατη λύση είναι οι ζωοτροφές, μα εδώ εμείς απαγορεύσαμε να δίνονται υπολείμματα κουζίνας και διάφορα ζουμιά περίεργα σε ζώα. Ε, θα πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη ειλικρίνεια όταν αποφασίζουμε αυτά τα θέματα. Γορέσαμε το χυλό, θυμάστε. Τώρα, αν μπορεί κανείς να φάει ένα γιαούρτι ή το προχθεσινό ξερό ψωμί, ε, δεν ξέρω το, αν θα πρέπει να τα συζητάμε εδώ. Ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι καταστρέφονται τρόφιμα. Σε αυτή εδώ την Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτούμε και ότι τα περισσότερα που, ε, ε, αυτό που επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον είναι η παρασκευή των τροφίμων, η ωραία συσκευασία, η ωραία παρουσίαση, το ωραίο το μιλαράκι που είναι καλά τυλιγμένο και μετά το πετάμε γιατί είναι λίγο ζουλιγμένο και δεν μας αρέσει και δεν θέλουμε να το φάμε και ενώ έχει φτάσει μέχρι το κατάστημα και το αγοράζουμε για να το πετάξουμε, όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε πώς λειτουργεί η αλυσίδα παραγωγής. Και να μπουν σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Χόρστ Σνέλχαρτ. Για να δούμε. Ε, πώς θα πάει από οικιακά. Ναι, εγώ υποστηρίζω αυτά τα οικιακά και την οικιακή οικονομία που ανέφερε η κυρία Κλάς ε, έχει δίκιο. Και πραγματικά τα λέει από σε αυτά. Βεβαίως, ε, στα τρόφιμα δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Ε, δεν θέλω να κάνω προπαγάδα ότι θα πρέπει να κοστίζουν περισσότερα, αλλά θα πρέπει στην κοινή γνώμη να ενημερώσουμε καλύτερα τον κόσμο για να εκτιμά το τρόφιμο. Και εκεί χρειάζεται λίγο μεγαλύτερο σεβασμός και προσοχή. Ε, βλέπω και εγώ τη συζήτηση στην κοινή γνώμη. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Καλχάης Φλόρενς. Δηλαδή, έχουμε αναπτύξει τόσες διαδικασίες, τόσες ρυθμίσεις. Εδώ εμείς οι ίδιοι τα αποφασίσαμε. Όπου τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο ε, με διάφορους τρόπους. Με αποστήρωση, με παστερίωση. Αν μπορώ σήμερα το γάλα να το κρατήσω πάνω από δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η βιομηχανία μειώνει την ημερομηνία ανάλωσης ε, για να πουλάει περισσότερο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδεολογία. Βάλε μικρότερη ημερομηνία να περάσει δύο μέρες να το πετάξει να πάρει άλλο. Σε πολλές συζητήσεις εδώ περιορίζουμε ε, τις ημερομηνίες και τα μέσα που θα μπορούσαμε ε, να χρησιμοποιήσουμε για να διαρκούν περισσότερο τα τρόφιμα. Αυτό που είπε Κρίστα ισχύει. Στις πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες ορίσαμε και αγωνιζόμαστε με νύχια και με δόντια σαν τρελή να χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Εμείς τα ορίσαμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Καλύτερα τα πετάμε αυτά τα προϊόντα ή τα καίμε εντάξει, μπορούμε να κερδίσουμε ενέργεια. Αλλά οι χωματερές είναι πραγματικά ένα θέμα, είναι ε, μια υπόθεση πεπερασμένη που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε πια. Υπάρχει νομοθεσία μας αφενός, αλλά αφετέρου χρειάζεται δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, για την παραγωγή τους, για την αξιοποίησή τους, για την εκτίμησή τους και από το σχολείο να ξεκινάει. Και στο σχολείο ε, υπάρχει μάθημα υγιεινή διατροφή. Τα τελευταία χρόνια αποτύχαμε. Ακριβώς γιατί ήταν πιο φθηνά τα τρόφιμα, είναι πιο φθηνά να το πετάς και να αγοράζεις άλλα. Εγώ δεν θέλω να ε, υπερασπιστώ τα ακριβά τρόφιμα, γιατί μετά ο κόσμος που είναι φτωχός δεν θα μπορεί να αγοράζει τρόφιμα. Δεν θέλω να το πάμε εκεί στη συζήτηση, να κρυβίνουν τα τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία η Κάριν Κάντενμπαχ. Συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Σνέλχαρτ. Κρίμα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο, γιατί η συζήτηση είναι συζήτηση αρχή. Αυτό το πρόβλημα ε, ακριβώ έχει φέρει στην επιφάνεια όλα τα θέματα που μα απασχόλησαν στο παρελθόν. Είναι θέμα του περιβάλλοντο, είναι θέμα τι γεωργία έχουμε και τι γεωργία θέλουμε, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και επίση και ένα ζήτημα ε, οικονομικού κέρδου και για μένα τώρα ίσως δεν περιμένετε να τα ακούσετε από μένα, είναι συντηρητική αντιμετώπιση. Εγώ δεν θα το βάλω στην οικιακή οικονομία και στον νοικοκυριό, αλλά στο θέμα της υγιεινής διατροφής. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε σε κάποιους άλλους ε, όλα τα θέματα της διατροφής. Έχουμε τρελαθεί με τις ετικέτες. Ο κόσμος αν δεν ξέρει τι είναι αυτό το τρόφιμο, από τι αποτελείται, τι συστατικά έχει, πώς επηρεάζει το μεταβολισμό, τι να την κάνει την ωραία ετικέτα που είναι τόσο σπουδαία, αλλά είναι για λίγους. Γιατί από χρόνο σε χρόνο αυξάνει ο αριθμό των αδαών. Και ε, και υπάρχουν παιδιά που ε, φτιάχνουν μόνα τους στο σπίτι διάφορα γλυκά, ξέρω εγώ μάφινς, δεν ξέρουν τι είναι αυτό, αλλά τους αρέσει γιατί είναι ωραίο, είναι γλυκό και δεν ξέρουν τι περιέχει καν τα συστατικά. Θα πρέπει τα παιδιά ε, στο σπίτι να μαθαίνουν τι είναι τα τρόφιμα, τι είναι τα συστατικά, τι είναι το μαγείρεμα, να έχουμε και άλλη οργάνωση στην κοινωνία, άλλα ωράρια εργασία, να μαγειρεύουν στο σπίτι, να τρώνε στο σπίτι, να ξέρουν τι μαγειρεύουν. Αν βγάλουμε τώρα ένα πετραδάκι από τη νομοθεσία δεν θα βοηθήσει. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να είναι σε όλες τις πολιτικές. Held in all policies το λένε αυτό στα αγγλικά. Καλό θα ήταν για τις συζητήσεις αυτές να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητούν τα κόμματα ξεχωριστά. Όλη η Ευρώπη προς τα που θέλουμε να προχωρήσουμε, ακριβώς για να μην έχουμε τέτοια προβληματική. Τόνους ολόκληρους πετάμε στα σκουπίδια τρόφιμα, δεν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Κρήτον Ασένης. πρακτικό παράδειγμα. I Το ήλπιζα, αλλά όχι. Θα ήθελα και εγώ να συμβάλλω στη συζήτηση. Για ένα λόγο, σε αυτή την αίθουσα δεν είδα ποτέ τόση μεγάλη συμφωνία των κομμάτων επί Όλοι που μίλησαν έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα. Αυτό είναι μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι με αυτή την κρίση ότι καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά που παράγουμε. Είναι θέμα που αφορά τι γενναίες, το περιβάλλον, τη διατροφή. Άπτεται αναπτυξιακών πτυχών Άρα θα πρέπει, ήρθε η ώρα για να λυθεί και νομίζω ότι είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, λέει ο Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις προ την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Σαντάλ Μπούτσι είναι εδώ από την Γενική Διευθυνσάνκο και θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Χόσπακ που μας παρήχε υποστήριξη και όλα τα άλλα μέλη. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Απόδειξη. Πρόσφατα στον οδικό χάρτη για την αποδοτική χρήση των πόρων θεώρησε τα τρόφιμα, όχι μόνο τη ότι τα τρόφιμα είναι πόρος που πρέπει να τον σεβαστούμε και να μην τον σπατάλαμε. Τώρα, η ημερομηνία κατανάλωσης και η ημερομηνία λήξης είναι πολύ σημαντικά και στις πληροφορίες που πρέπει να χορηγούνται προς τους καταναλωτές, σε απόφαση που έλαβαν τα θεσμικά όργανα, διαφορά μεταξύ των δύο κατέστη σαφής και πρέπει να καταστεί σαφέστερη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο βιομηχανία. Διότι η ημερομηνία κατανάλωση είναι θέμα ποιότητα. Είναι για τα, για τα ζυμαρικά, για το ρύζι, ε, για τα δημητριακά και μπορεί να τα φας πολύ μετά από την ημερομηνία. Η βιομηχανία βάζει αυτή την ημερομηνία για να είναι σίγουρη ότι είναι ποιοτικό και νόστιμο το προϊόν, αλλά μπορεί να το φας και πολύ αργότερα μετά αυτή την ημερομηνία. Και δεν το ξέρουν όλοι οι καταναλωτές, πράγματι. Η άλλη ημερομηνία πολύ πιο σημαντική διότι αφορά θέματα υγείας, ασφαλείας και η ημερομηνία λήξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ημερομηνία μέχρι πότε μπορεί να απολύεται το πρόβλημα. Εκεί το πώς καθορίζει η βιομηχανία την ημερομηνία λήξη υπάρχει περιθώριο λιγμών. Ποσοστό ασφαλείας. Υψηλότερο ποσοστό, χαμηλότερο ποσοστό ασφαλείας για τα γιαούρτια. Για να είναι ασφαλής δίνουν μια ημερομηνία που είναι αυστηρότερη, για άλλα προϊόντα είναι πιο χαλαρή. Αλλά σχετίζεται με την ασφάλεια μικρο, ε, μικροβιολογική ασφάλεια κλπ. Κάποιοι αναφέρθηκαν στη συσκευασία. Σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά μέχρι κάποιο βαθμό βέβαια. Διότι η συσκευασία πρέπει να βελτιστοποιείται και δεν θα πρέπει να αυξάνεται. Αν πρέπει να συσκευάσεις τα πάντα για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, τότε έχει και περισσότερε συσκευασίε που πρέπει να πάνε στη χωματέρη. Άρα χρειάζεται βελτιστοποίηση τη συσκευασία. Καμιά φορά με σακούλες που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, καμιά φορά συσκευάζοντα μικρότερε δόσει. Και εδώ υπάρχουν δυνατότητε για έρευνα και για καινοτομία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αναφέρθηκε η νανοτεχνολογία σαν παράδειγμα. Θα πρέπει όμω να έχουμε να εξετάσουμε την ασφάλεια και πώ το δέχονται οι καταναλωτέ. Μπορεί να δεχτεί ο καταναλωτή να έχει συσκευασία που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την κατάσταση του φαγητού, του τρόφιμου. Αυτό εξετάζεται ακόμα. Κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι οι φορεί τη τροφική αλυσίδα πρέπει να παίξουν τον ρόλο του από τη γεωργία μέχρι τον καταναλωτή. Στατηγική των λιανοπολιτών αναφέρθηκε αυτή επανειλημμένα. Ε, είναι πολύ ανταγωνιστικό τομέα. Συχνά ακολουθούν κάποιε στατικικέ για να γεμάτα τα ράφια όσο γίνεται. Σε κάποιε περιπτώσεις πρέπει βέβαια όμω να αδειάζουν τα ράφια διότι έχουν ε, παλιώσει κάποια προϊόντα και δεν έχουν πολιθεί. Και πολύ συχνά και η εικόνα των λαχανικών επιβάλλεται από του και από του πελάτες. Ένα καρότο που είναι στραβό το πετάνε το χάρη. όταν τα μαζεύουν και το χωράφι. Διότι δεν είναι τέλεια ίσιο το κάροτο. Καμιά φορά το παίρνουν για άλλη χρήση, αλλά πολύ συχνά τα αφήνουν στο χωράφι και το μαζεύουν το κάροτο. Ε, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ε, βιομάζα το απορριπτόμενο τροφίμο. Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή την πολιτική. Δηλαδή, να το κάνουν επιχείρηση οι εταιρείε. Να έχουν δηλαδή να πετυχαίνουν, να έχουν δυνατόν περισσότερε απορρίψει τροφίμων να τα χρησιμοποιούν για βιομάζα. Στην Νότια Αγγλία Υπάρχουν εταιρείε που μαζεύουν ξεχωριστά τα απορρίμματα των τροφίμων ε, για βιομάζα. Όταν αυτό δεν αποφευθεί είναι καλό. Δεν έχουμε ένα αρμονισμένο σύστημα με δεδομένα στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι γίνεται στον οικοκυριό, πόσα τρόφιμα απαιτιούνται. Καθημερινά ζυγίζονται οι συλλογή στοιχείων σε μεγάλη αγορά των Παρισίων που είναι κεντρικός κόμβος για διανομή των τροφίμων μας είπαν ότι καθημερινά πετάγονται 8 τόνοι νοπών τροφίμων. Όχι γιατί σέβεται ο κόσμος τα τρόφιμα, είναι θέμα οργάνωσης. Είναι λιγότερο πανηρό να πετάξουν τα τρόφιμα παρά να έχουν σύστημα μεταφοράς αυτών για να φτάσουν τα τρόφιμα είτε στους καταναλωτές είτε σε καταστήματα τροφίμων ή σε άλλους διανομής. Άρα το όλο σύστημα πιθανότατα χρειάζεται επικαιροποίηση εν γέννη. Έχουμε την εντύπωση ότι όλοι συμφωνούμε με το στόχο. Πρέπει να δούμε πώς το πετύχουμε καλύτερα όμως. Είναι θέμα συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων. Είναι θέμα πιθανότατα τεχνολογίας, επιμελητίας, μεταφοράς. Και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Και έχω υπόψη μου λέγοντας αυτό τα κάτι μέλη, την τοπική αυτοδίκηση στη συλλογή των ε, απορριμμάτων πραγματος χάρη. Πρέπει να δούμε πού γίνεται η μεγαλύτερη σπατάλη. Εμείς νομίζουμε σε, όλη της, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του καταναλωτού, να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι συμφωνούμε με τους βασικούς στόχους να αποφευθεί πρώτα απ' όλα και όταν δεν μπορεί να αποφευθεί να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτών των απορριμμάτων. Ελπίζω να ακάλυψα τι ερωτήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχει σχετική συνένεση ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και ότι η στρατηγική, αναφέρθηκε μάλλον και η στρατηγική της ε, αποδοτικότητας ε, των πόρων και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε πού μπορούμε να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί. Ιδάλλως δεν θα πετύχουμε τις στόχους μας. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την Άννα Ασπακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα είναι πάρα πολύ θετικό να ακούμε τι λένε και οι συνάδελφοι και είναι πάρα πολύ καλό πάντα όταν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Φυσικά μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση. Στην γνωμοδότηση. Γίνεται λόγος για τα βιοκάψιμα στην ε, έκθεση. Ασφαλώς επειδή πρόκειται για ζητήματα που μπορεί να υπάρξει εκ νέου αξιοποίηση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα αυτά, γιατί για παράδειγμα περιέχουν πολλή υγρασία και προαπαιτούν μεγάλη ενέργεια, μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να επαναχρησιμοποιηθούν ως βιομάζα, ως βιοκαύσιμα. Άκουσα αυτά που είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι. Είναι καλή ιδέα θεωρώ σε κάποια φάση να θέσουμε τους δικούς μας κανόνες για τα τρόφιμα. Πολύ σωστές οι ιδέες των συναδέλφων. Το θέμα είναι ουσιαστικά ότι έχουμε υπερβολικούς, πολλού, υπερβολικά πολλούς και αντιφατικούς νόμους. Στην Δανία, στη χώρα μου παλιότερα, είχαμε δύο πληροφορίες για τα τρόφιμα. Μέχρι πότε το τρόφιμο μπορούσε να παραμείνει στο σούπερ μάρκετ, στα ράφια και μια ημερομηνία για την ε, κατανάλωση, για τον καταναλωτή. Μέχρι πότε μπορεί να καταναλωθεί ένα προϊόν. Αυτά λόγω Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καταργήθηκαν. Θα δούμε πώς πρέπει να τα επανεισάγουμε. Άλλο ένα πρόβλημα έχω σε ό,τι αφορά τι συσκευασίε. Ήμουν πρόσφατα, πήγα στο Βερολίνο, μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ λοιπόν και διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι υπήρχαν διάφορα φρέσκα προϊόντα τα οποία μπορούσε να τα αγορέσει... κανένας ε, σε, μεμονωμένα. Γιατί και εγώ μένω μόνη και τα χρειάζομαι μεγάλες συσκευασίε. Συμφωνώ λοιπόν με την τάση αυτή. Και είναι άλλωστε παράλογο να χρησιμοποιείτε και τόσο πολύ ε, πλαστικό για τη συσκευασία. Καλό θα ήταν ίσως να αγοράζονται έτσι σκέτα τα προϊόντα. Τα οποία να τα παίρνει κανείς όπως θέλει, ό,τι ποσότητα θέλει και να τα βάζει στη σακούλα του. Κάτι άλλο τώρα. Για τα κατεψυγμένα προϊόντα. για, ε, για τα μικρά νοικοκυριά μπορεί και αυτά να κάνουν τη διαφορά. Γιατί μπορεί κανείς να βγάλει ό,τι ποσότητα θέλει και το υπόλοιπο να το κρατήσει στην κατάψυξη. Όλοι θεωρούμε ότι το θέμα αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όλο και πιο πολλοί κόσμος δεν έχει να φάει στον κόσμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η ιδέα. Η συζήτηση η οποία ήταν πάρα πολύ ε, καρποφόρα σε ό,τι αφορά τις ιδέες που ακούσαμε και 19 Οκτωβρίου στι 12 ε, είναι η προθεσμία κατάλυσης τροπολογιών, 22 Οκτωβρίου ε, ψηφίσουμε. Η Επιτροπή Γεωργία θα ψηφίσει στις 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να πάρει υπόψη και τη γνωμοδότησή μας. Συνάδελφοι, <laughs> δεν έχει ακόμα καταφτάσει το αεροπλάνο από την Κοπεχάγη, άρα τι να κάνουμε. Ε, α, α, μα, μα, μα συγγνώμη, έφτασε το αεροπλάνο. Μα ήσασταν πάρα πολύ διακριτικοί. Χωρίς θόρυβο και χωρίς... Ε, εκπομπές ε, αερίων. Ήρθε το αεροπλάνο λοιπόν στην αίθουσα, άρα να δούμε πρώτα το σημείο 3 της σημερινής διάταξης. Καλώς ορίσατε. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Άρα, θα περάσουμε τώρα στο σημείο 3 της σημερινής διάταξης. ορίζουμε, λοιπόν την Τζακλίν Μαγκλέιρ, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος από την Κομπεχάγη. Καλώς ορίσατε στην τακτική ανταλλαγή απόψεων, την οποία διεξάγουμε εδώ μαζί σας στην Επιτροπή μας, να ακούσουμε τι έχει συμβεί το 2011 και ποια project βρίσκονται προθυρών. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ακούσουμε πολλά. Υπήρξε και μία αποστολή στην Κοπεχάγη στις αρχές Σεπτεμβρίου και οι συνάδελφοι θα μας αναφέρουν τα όσα είδαν. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο να μας κάνετε την παρουσίαση των εργασιών σας. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη άφηξη. Τα κατάφερα μέσω μονάχου και επικοινωτρόπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου διαθέτετε χρόνο να σας μιλήσω για το έργο του οργανισμού, τι κάναμε το 2011 και το πρόγραμμα εργασιών για το 2012. Βέβαιως συνεχίσαμε να κινούμεθα σε ευρύ πεδίο πολιτικών προσπαθώντας να υποστηρίξουμε τις διάφορες ζητήσει που, που διέπονται από τον δικό χάρτη για την αποδοτική χρήση των πόρων. Θέλαμε να πετύσουμε βιοκυλότητα, προστατεία προστασία των υδάτων, της γης, ενέργεια, κλίμα κλπ. Να τα καλύψουμε όλα αυτά. Το 2011 τονίσαμε εκ νέου, στη συνεργασία με το δίκτυο και με τα κράτη-μέλη, τονίσαμε λέγω ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμεθα και εργαζόμεθα. Θα πρέπει να γίνουμε αποδοτικότεροι στη συλλογή πληροφοριών, τη μεταβίβαση πληροφοριών και να προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ πιο καλά ενημερωμένοι με πρόσφατες πληροφορίες και να κινούμεθα έγκαιρα. Όσον αφορά το κοινό σύστημα πληροφοριών για το περιβάλλον, θα σα ενημερώσω και πώ βοηθούμε χώρε να, διάφορες, να υιοθετούν διάφορε αρχέ υπέρ του περιβάλλοντο προτεραιότητες το 2012 έχουν βασιστεί το 2011 ο οδικός χάρτης, εμποτική χρήση των πόρων, πράσινη οικονομία, λογιστική του οικολογικού συστήματος, ε, για μείωση της, των αλλαγών του κλίματος, ε, επιμερισμός των προσπαθειών, θέματα προσαρμογής. Θα έπρεπε να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ε, ετοιμάζουν τις εκθέσεις τους και την ενημέρωση και να παράσχουμε υποστήριξη μέσω συζητήσεων περιδικτών ούτω ώστε να δούμε ποιε επιδοτήσει είναι επιβλαβεί το περιβάλλον και ποιε φορολογικέ μεταρρυθμίσει χρειάζονται και να δούμε πώ μπορούν να κινηθούν οι χώρε και πώ μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά του όσον αφορά του πόρου που χρησιμοποιούν. Εν συντομία λοιπόν, έχουμε παράγει διάφορε εκθέσει. Να σα δώσω κάποια ιδέα. Τι τελευταίε εβδομάδε μόλι ε, ε, υποβάλαμε σημαντικά πορίσματα για το θέμα της αλλαγής του κλίματος, για, για τις τάσεις και προβολές για το εθεμοκηπείο 2011, αναδρομική ανάλυση, 20 χρόνια ε, δραστηριότητάς μας, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, βρήκαμε τρόπο να εκτιμούμε ποια θα είναι η μορφή των διαφόρων καταγραφών των, στοιχείων των ε, χωρών ένα χρόνο πριν από αυτά που βλέπει ο ΙΕ για την αλλαγή του κλίματος και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις μας είναι εντό των ορίων ε, των, των προβλέψεων. Μεγάλη έκθεση για την αποδοτική χρήση των πόρων. Βλέπουμε πώ οι διάφορε χώρε προσεγγίζουν το θέμα και μετά σε δύο εβδομάδε θα ξεκινήσει η έκθεση για τι μεταφορέ και το περιβάλλον. Θα υποβάλουμε το πορίσμα, την έκθεσή μα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά θα ετοιμάσουμε έκθεση για την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Εξακολουθούν να εκπονούνται εκθέσεις. Τι μας λένε ότι σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούμε να είμαστε μακριά από τους περιβαλλοντικούς μας στόχους όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Είμαστε καθοδόν προς τις υποχρεώσεις του Κιώτο, αλλά είχαμε αύξηση το 2010 περίπου 2,4%. Το 2009 είχαν μειωθεί οι εκπομπές και αυτό ακυρώνει κάπως την αύξηση, άρα είμαστε ακόμα εντός των στόχων Αυστρία, Ιταλία και Λουξεμβούργο πρέπει να κινηθούν. Πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα όσον αφορά του εταιρικού του μηχανισμού και τι πολιτικέ για να συμμορφωθούν. Τώρα για το 2012, στο μέλλον, θέλω να δούμε ποια οικοδομικά στοιχεία θα αλλάξουν, αν θέλετε. Θα εστιαστώ πρώτα απ' όλα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη νέα δουλειά που θα αναλάβουμε όσον αφορά τις εκπομπές και τον επιμερισμό των προσπαθειών. Τα αποτελέσματα που εισέφθηκαν πρόσφατα μας δείχνουν τι θα γίνει μέχρι το 2012. Μετά από αυτό εσωτερικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επεξεργαστεί τον ορισμό των ετησίων νομών και εκπομπών κάθε χρόνο για να πορεύονται τα κράτη-μέλη. Είναι βασικό κεντρικό σημείο αλλά και επίμαχο με διάφορες χώρες. Και ο οργανισμό θα είναι διαφορετική θέση από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν εξ αυτού. Πρωταρχικά διότι όχι μόνο θα εξετάζουμε και τα τμήματα, τα εμπορεύσιμα της οικονομίας και τα μη εμπορεύσιμα. Άρα μέσω γραμματείας θα γίνει εξέταση πλευράς εμπειρογνωμών σε κάθε χώρα για να δούμε τι θα κάνουν σε εθνικό επίπεδο και τα συμπεριλάβουν στο εθνικό τους απολογισμό. Πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε ξαναθέσει προτεραιότητες στον φωτοπροσωπικό. Βασική αλλαγή είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε εμπειρογνώμονες που είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς. Να συμμετέχουν σε μία ομάδα που θα μετακινείται και θα εξετάζει τι γίνεται στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη και τι γίνεται με αυτές τις απογραφές τους. Και αυτό θα έχει μεγάλες ε, οικονομικές συνέπειες όσον αφορά την ποδική χρήση των πόρων. Συνεργαστήκαμε πολλούς συναδέλφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και μέσα στο Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει, τι θα φέρει το μέλλον όσον αφορά μελλοντικού υπολογισμού των ερευνών για την ετήσια ανάπτυξη. Και ελπίζουμε ότι εντός ενός έτους θα δώσουμε πιο επίσημη χρειά στον απολογισμό των στοιχείων ενεργητικού της, ε, ενεργητικού της Ευρώπης. Προσημοποιούμε τη γη, τον άνθρακα, το νερό, τον άνθρακα ιδιαίτερα. Και αυτά ακολουθούν αυτά που έχουμε ήδη στη χέρια μας τώρα όσον αφορά την ε, εσωτερική κατανάλωση. Συνεργαζόμαστε και με τον ΟΗΕ, στα στατιστική υπηρεσία του ΟΗΕ και με την Παγκόσμια Τράπεζα και ελπίζουμε το 2012 οι εργασίε αυτέ αναγνωριστούν διεθνώ ω προσεγγίσει και να χρησιμοποιηθούν παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη. Όσον αφορά βιοπικιλότητα και νερό, δεν θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε την υφιστάμενη νομοθεσία για τους βιοτόπους, για τα πτηνά και τη Ανατούρα 2000, αλλά να επεκταθούμε και στην πράσινη υποδομή. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε ποια θα είναι η βάση αναφοράς και οι σχετικοί χάρτες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τι συνέπειες έχουν οι μεταφορές και οι άλλοι τομείς στην πράσινη υποδομή της Ευρώπης, πέραν αυτού. Θα επεξεργαστούμε την αξιολόγηση των οικοσυστημάτων μαζί με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και θα εξετάσουμε και τη Σύμβαση για την της Ναγκόγια. Του νέου στόχου. για να δούμε πώ θα του πετύχουμε. Και για τη μέτρηση και την υποβολή αναφορών και την εφαρμογή των μέτρων. Διεθνώ θα υποστηρίζουμε το μηχανισμό του συμψηφισμού, clearing house, και ελπίζουμε να κινητοποιηθούν και άλλε χώρε αντίστοιχα, και η κοινωνία των πολιτών και κυβερνήσει. Και για τη βιοποικιλότητα, αλλά για συνέπειε αλλαγή του κλίματο και για τα μέτρα προσαρμογή σε αυτέ τι αλλαγέ. Τώρα, πώ κινούμεθα για τη βιοπικιλότητα, να σα δώσω μια γεύση. Στο Ρίο Προσπαθούμε να δείξουμε γιατί είναι το σημαντική βιοπικιλότητα. Μέσω κατανόησης των τροφίμων. Και συζήτησαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάνω σε αυτό. Και τι βλέπουμε. Κάποιοι από καλύτερους τη βιοπικιλότητας προέρχονται εκτός από τον κόσμο της συντήρησης από αρχιμαγείρους και άλλους που υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η βιοπικιλότητα για να φτιάξουν τα φαγητά τους. Στο Ρίο Συν θα αναλάβουμε να ετοιμάσουμε μια εκδήλωση, μεγάλη εκδήλωση, με πολλού συναδέλφου από όλο τον κόσμο, να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτήν την ιδέα τη βιοπικιλότητα. και το τι βλέπουμε στις ε, τοπικές κουζίνες και στη δίαιτα. άλλο ακρογωνίο λήθος για το Ρίο Συν 20, βάσει της δημιουργική στην Αστάνα που μόλι έλαβε χώρα, είναι η παγκόσμια αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινού συστήματο περιβαλλοντικών πληροφοριών που είχαμε στην Ευρώπη και ακριβεί αρχέ. Αυτέ οι ακριβεί αρχέ γρήγορα γίνονται σημαντικότατο ακρογωνέ λήθος όσον αφορά την παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Τόσο πολύ που πιστεύω ότι τελικά πιθανότατα κάποια τμήματα θα εμφανιστούν εντό ε, των δηλώσεων του Ρίο. Ε, διακηρύξεων του Ρίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τρόπο συνεργασία με διάφορέ χώρε. Πέρα από τη σύμβαση του Άρχου. Και έτσι θα καταλήξουμε σε πιο ανοιχτή εκτίμηση ε, των μεθόδων επαλήθευσης, ελέγχου, υποβολής αναφορών. Αυτό το έργο μας υποστηρίχθηκε από την ΤΕΦΚΟ, γειτονία στην πολιτική γειτονίαση προς Ανατολάς και προς Νότον. Πολύ προσοχή προσδίδεται και ενδιαφέρον υπάρχει σε χώρες που συνεργάζονται μαζί μας όσον αφορά αυτές τις αρχές από Ρωσία μέχρι την Ισία. Μία από τις δυσκολίες που προβλέπουμε όμως που διαφαίνεται είναι το GMS e θα πρέπει να είναι εκτός του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό δημιουργεί προβλήματα για πολλά πράγματα που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε εντός της Ευρώπης. Το είχαμε προβλέψει τι θα κάνει το GMES για τη δική μας δουλειά, για τη δική μας ανάπτυξη των διαφόρων υπηρεσιών όσον αφορά τη γη και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την επισκόπηση μας των δορυφόρων ε, για τους σκοπούς μας και χρειάζεται τεράστια επένδυση, 2,3 δις ευρώ που ήδη έχουν διατεθεί. Τι βλέπουμε, ότι χωρίς το GMS, e εάν δεν ήταν εντός δημοσιονομικού αυτού πλαισίου, αν δεν θα υπάρξει πραγματικό πρόβλημα υποστήριξη τη γεωργίας, του τρόπου με τον οποίο θέλουμε να περιγράψουμε τη χρήση των γεών, την αλλαγή χρήσεω γεών, τη λογιστική όσον αφορά τον άνθρακα κλπ. Ένα αίτημα θα είχα να σα υποβάλω, να επανέλθουμε ξανά στο GMES και να δούμε πόσο σημαντικό είναι για πάρα πολλέ από τι ε, πολιτικέ που ενδιαφέρουν και την Επιτροπή σα, αλλά και πολλέ άλλε, θα έλεγα. Θαλάσσια πολιτική, μεταφορέ, γεωργία, περιφερειακή ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Εν κατακλείδη, ήθελα να πω ότι βεβαίω είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, θέλουμε να σα υποστηρίξουμε ε, όσον αφορά την ανάπτυξη του 7 πλαισίου, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είπαν ότι θα πρέπει να είναι έτοιμο αυτό το πλαίσιο ε, τον Ιανουάριο, δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή όχι, αλλά το υποστηρίζουμε. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τι ανάγκε σα και ήδη προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό όχι μόνο τη ε, εκθέσεω για την κατάσταση του περιβάλλοντο, αλλά θέλαμε να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε από χώρε και τα κράτη-μέλη να δουν πώ θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα εφαρμογή. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε διάλογο με διάφορες χώρες για να ξεκινήσουν πιλωτικές μελέτες στους τομείς των αποβλήτων και την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα και ενδεχομένω και στη βιοπικιλότητα για να διερευνήσουμε πραγματικά πέρα από τον αυστηρό τομέα της συμμόρφωσης, δηλαδή την εσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία, να δούμε γιατί η νομοθεσία και διάφοροι τομείς πολιτικής υποφέρουν από κακή εφαρμογή. Αυτό μπορεί να είναι μη συμμόρφωση, μπορεί να οφείλεται σε πολλά άλλα θέματα, έλλειψη επενδύσεων κλπ. Οπότε μαζί με το δίκτυο EPA έχουμε ήδη εντοπίσει διάφορες χώρες για το 2012 όπου θα εξετάσουμε τι γίνεται με τα πόβλητα και σπατάλη και όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας θα συνεργαστούμε με πόλεις για να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να πετύχουμε την πλήρη εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών που συζητούμε. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα σταματήσω κάπου εδώ και με τα χαράς βεβαίως να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που αφορά και το πρόγραμμα εργασιών για τον επόμενο χρόνο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλέιτ για αυτή την επισκόπηση που μας δώσατε. Οι διερμηνείς θα χρειαστεί να πάρουν μια βαθιά ανάσα μετά από όλα αυτά. Όντως, θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι για πολλούς τομείς ε, η βάση για καλή πολιτική είναι τα καλά στοιχεία και η ενημέρωση από δορυφόρους είναι πραγματικά ε, ζωτική σημασία παρευρίσκεται η Γιώτα και η συγγήτρια για τον προπολογισμό και μάλλον ε, θα έχει κάτι να μας πει για το πώς θα εξασφαλίσουμε αυτό το σύστημα GMES που είναι η Παγκόσμια Παρακολούθηση Περιβάλλοντος και Ασφάλειας, ε, να εδραιωθεί στον προπολογισμό και να μην είναι έτσι κάτι το παροδικό, αλλά να παραμείνει. Έβδομο πρόγραμμα δράσεις για το 2012 για το περιβάλλον και φαντάζομαι και ο Οργανισμός Περιβάλλοντος θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα που μας ε, απασχολεί πάρα πολύ είναι ο παράγων Ε, των βιοκαυσίμων. Δηλαδή, ε, με τα βιοκαύσιμα μήπως τελικά κάνουμε ζημιά, γιατί ε, αφιερώνεται η γη σε άλλους σκοπούς, δεν ξέρω τι αποτελέσματα έχουμε. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τα ευρήματά σας. Έχουμε και ένα σύνδεσμο με τον οργανισμό σας, που είναι ο κύριος Γκερπράντη και του δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μακλέιτ και πάλι για την παρουσίασή της, ήταν πολύ σαφής. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, θερμότατη υποδοχή που μας επιφυλάξετε πριν από λίγες εβδομάδες όταν ε, μετέβημε με αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στον οργανισμό σας. Το συζητήσαμε για αυτό το θέμα της επίσκεψης πριν από δύο εβδομάδες περίπου στην Επιτροπή εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η μία αφορά τα απόβλητα η πολιτική τον έχει τεράστιο πρόβλημα στην εφαρμογή της, όπως είπατε. Μιλήστε για μερικά πιλωτικά προγράμματα. Σκέφτεστε ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει κανέναν άλλο ρόλο ο οργανισμός σας με την υποστήριξη, ακόμα και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρατών μελών στην υλοποίηση της νομοθετίας περί αποβλήτων, ιδιαίτερα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Uh, under pressure Για ε, βιοπικιλότητα. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης πίεσης. Βλέπετε διάφορα γεγονότα μη αντιστρέψιμα. Ίσως ε, να εμπνέομαι από τη χώρα μου ε, βλέπω ε, πολιτικούς και υπουργούς να διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τους στόχους που βάζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και παρόλο που διαφωνούν ε, κάποιοι επιστήμονες, ο υπουργός λέει ότι θα φτάσει στους στόχους, αλλά ε, αν γίνει αυτό κάποια στιγμή ο ίδιος θα έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό και δεν θα μπορεί να αποδείξει τίποτα. Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο εκεί ο οργανισμός σας, γιατί μιλούμε για πολιτικές που θα έχουν αποτέλεσμα σε 10-15 χρόνια. Δεν ξέρω, ίσως εσείς μπορείτε να μας, το απαντήσετε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Γκερμπράντη. Υπόλοιποι ομιλητέ, ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω κύριε ε, Γενική Διευθύντρια να πω δύο λόγια. Αν κοιτάξουμε τον προπολογισμό που κατατέθηκε τις τελευταίες μέρες, νομίζω μπορούμε να είμαστε περήφανοι που έχουν μπει στον προπολογισμό τόσα στοιχεία για την βιωσιμότητα και την αηφορία. Θα με ενδιέφερε να ακούσω το ρόλο που διαδραματίζει ο δικός σας οργανισμός, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και στατιστικών που είναι τόσο σημαντική. Πώς συνεργάζεστε εσείς με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές. Γιατί συζητήσαμε και τους συνολικούς λογαριασμούς που λαμβάνουν υπόψη και το περιβάλλον στα οικονομικά. Όλα αυτά λειτουργούν. Η συνεργασία πώς έχει με τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές. Ε, τι γίνεται με την ανταλλαγή στοιχείων στατιστικών για να έχουμε μια ασφαλή βάση δεδομένων και αξιόπιστη. Και την τελευταία φορά συζητήσαμε αυτά τα στοιχεία, αλλά τι θα γίνει με τη διάδοση, γιατί γνωρίζετε ότι η πολιτική ζει και από την ενημέρωση της κοινή γνώμη. Και σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά στοιχεία έχω την εντύπωση ότι δεν ε, διαδίδονται αρκετά. Μερικά είναι ανισχυτικά, αλλά δεν είναι γνωστά η δική σας υπηρεσία, ο δικός οργανισμός πώς μπορεί να συνεισφέρει. Και μια τεχνική ερώτηση. Αναφερθήκατε για, στην ποιότητα του αέρα. Θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια για τα ορούμενα σωματίδια σκόνης. Γιατί σε πολλές χώρες συμβαίνει αυτό, ε, ξεπερνούν τα όρια. Ε, ποια είναι η στατιστική βάση για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Chris Davis. Να συνεχίσω πάνω σε ένα-δύο θέματα που με ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα ανταλλαγής ρήπων και στόχους μειώσεως διοξιδίου του άνθρακα. Αναφέρεται την Ιταλία. Η Ιταλία ότι ήταν εκτός στόχων. Αυτό δεν υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα. Μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω. Όσον αφορά στόχους του 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα θυμίζει ότι όταν οι πολιτικέ εφαρμοστούν πλήρω, να φτάσουμε σε μείωση 25% όσον αφορά τα νοικοκυριά μέχρι το 2020. Με, εσωτερικά μέσα μάλλον το 2020. Αποδοτική, αποδοτικότητα για την ενέργεια είμαστε μακριά. Το 3% ανάπτυξη, αύξηση των εκπομπών πέρσι. Και εξακολουθείτε να λέτε είμαστε στο στόχο του 2020 και εγώ βλέπω το 3% και μου δημιουργείται ένα ερωτηματικό στο μυαλό βλέποντας την τιμή του άνθρακα σήμερα και την ανεπάρκεια του συστήματος εμπορίου α, ρήπων για την εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση σε άνθρακα. Και έχω ερωτηματικό και στον αφορά αυτό το στόχο. Πόσο κινδυνεύουμε να χάσουμε το στόχο. Ένα στόχο που είχαμε συνηθίσει να τον θεωρούμε σαν σίγουρο. Μαργαρίτα Αουκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. λέει η κυρία Άουκεν. Η τελευταία συνάντηση στην Κοπενχάγη ήταν πολύ χρήσιμη και θα το συνδέσω με το θέμα της βιομάζας και την αλλαγή του κλίματος. Η ουδετερότητα του κλίματος, η υπόθεση για μηδενικές εκπομπές, μέσω χρήσεως βιοκαυσίμων για ενέργεια. δεν δικαιολογείται αυτό το μέσο σαν ουδέτερο, για να το πω ήπια. Μετά, μπορείτε να αναλύσετε περισσότερο. Τι, με τις ζωοτροφές πώς επηρεάζουν, με τον κύκλο των ζωοτροφών και τα απόβλητα της ζωοτροφές πώς επηρεάζουν το κλίμα. Διάφορες πηγές ε, κατάλοιπα, ε, ξυλία κλπ. Κάνατε έξοχη δουλειά ξεκαθαρίζοντας πόσο πολύτιμο, πολύτιμα μπάνε τα απόλυτα, είναι πόρος. Θεωρείται όμως ο φυής τρόπος χρήσεως αυτού η καύση. Μπορείτε να μας δώσετε ακριβή στοιχεία. Τέλος βιωσιμότητα, κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα θα ήταν χρήσιμο συσχετιστούν με τη... Ούτως, να έχουμε σαφή στοιχεία να μπορούμε να κάνουμε συσχετισμού για να υπάρχουν και συγκεκριμένε προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κυρία Διευθύντρια για την παρουσίασή σα αλλά και για το έργο που επιτελείτε στον οργανισμό σα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον πρόεδρο Λάινεν και τον Κρίς Ντέιβις Ω προ τη σχέση τη αξιολόγηση με την πολιτική. Αν θέλουμε πραγματικά να βαρύνουμε με τα επιχειρήματά μας θα πρέπει αυτά να είναι οικονομικής φύσεως. Αλλά η αξιολόγηση που κάνετε εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για μας από την ποσοτική αξιολόγηση θα πρέπει να περάσουμε στο κόστος ε, αντιμετώπισης και σε, να συγκρίνουμε το κόστος πρόληψης και να δείξουμε πόσο η πολιτική πρόληψη ανεξάρτητα από το περιβαλλοντικό ας πούμε στοιχείο τα θέματα πρόληψης είναι ενδιαφέροντα και από πλευράς οικονομικής και συμφέρουν. Ε, πραγματικά έχουμε ανάγκη κάτι τέτοιο και με τις δικές σας αξιολογήσεις μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό. Το θέμα τώρα της εξωτερικεύσης είναι πραγματικά κομβικό, είτε το λέμε είτε όχι, όταν γίνεται λόγος για ε, το φόρο διοξιδίου του άνθρακα, τη μονάδα ε, βιοπικιλότητας κτλ. Όλα αυτά είναι εξωτερικά στοιχεία, αλλά προχωρούμε πάρα πολύ αργά σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε του χρόνου να έχουμε μια πρώτη έτσι, λογιστική εκτίμηση των πόρων. Ε, πώς μπορούμε δηλαδή ε, λίγο να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία για να περάσουμε πιο γρήγορα από τα ποσοτικά στοιχεία στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και έτσι να στοιχειοθετήσουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις προτάσεις της Επιτροπής μας, που συχνά είναι αντικείμενο παρανόησης από μέλη άλλων επιτροπών, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, γιατί δεν βλέπουν το οικονομικό όφελο. σε πάση περιπτώσει. Αναφερθήκατε στο θέμα της ποιότητας της ατμόσφαιρας του αέρα και έχετε εισάγει και διάφορα μέτρα, το ανέφερε και ο συνάδελφος Ζέμπερ και έθεσε σχετική ερώτηση όλο και πιο πολλά αυτοκίνητα diesel ε, κυκλοφορούν στα αυτοκίνητα, αλλά ε, προσθέσαμε και το NOx στα του αζότου στα, στις ουσίες αυτές που μετράνε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιφατικό αυτό. Μήπως χρειάζεται μια στρατηγική από πλευρά ε, του οργανισμού για το περιβάλλον, για το τι θα κάνουμε στο μέλλον, γιατί επίκειται και διάφορες αναθεωρήσεις και κάποια στιγμή ως νομοθέτες θα πρέπει πέρα από πρότυπα να δίνουμε και τα απαραίτητα μέσα για να πετυχαίνουμε αυτά τα πρότυπα. Τη δική σας άποψη θα ήθελα να ακούσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος, κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχαμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Περιβάλλον και για τον ενθουσιασμό που σας διακατέχει. Αυτή ήταν τουλάχιστον η δική μου εντύπωση. Όπως και οι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να κάνετε ακόμη πιο πολλές αναλύσεις. Έριξα πριν από λίγο μία ματιά για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιπληχθεί από τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά ανθρώπους που αρρωσταίνουν. Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Τι γίνεται με τα χημικά, για παράδειγμα, και μιλώ κυρίως για τις ε, χώρες προσανατολάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις ή μόνο συστάσεις. Μπορούμε να κάνουμε επίσης μια άλλη παρόμοια ερώτηση σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της ποιότητας των υδάτων στην Ευρώπη. Πόση μόλυνση υπάρχει, πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και με ανησυχεί ιδιαίτερα στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρος. Πολλές ερωτήσεις. Να ακούσουμε και τις απαντήσεις τώρα. Να προσπαθήσω, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα απόβλητα και η ποιότητα των ε, υδάτων και η βιοποικιλότητα αποτελούν τον πυρήνα των εργασιών μας ακόμη. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τα κράτη-μέλη για να περάσουν πέρα από την φάση της εφαρμογής της νομοθεσίας, να μας δώσουν πιο πολλές πληροφορίες για τις βιωτικές συνθήκες των πολιτών τους. Δεν θέλω να προκαταβάλω την έκθεση που θα δημοσιευθεί από τον οργανισμό μας σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες, θα ήθελα να πω ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουν ε, ε, δημοσιεύσει τα κρατημέλη στο EPR και στο ETR και έχουμε κάνει μια οικονομική ανάλυση των στοιχείων αυτών. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο και πιο πολύ να σας δώσουμε ως Επιτροπή και σε άλλες Επιτροπές τα μέσα εκείνα, τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία ήταν πραγματικά καταδεικνύουν γιατί δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις προσπάθειές μας. Αντιθέτως θα πρέπει να τις εντείνουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, αλλά και σε ό,τι αφορά άλλα θέματα. Όπως όσον αναπτύσσεται η επιστήμη, διαπιστώνουμε ότι είναι θέμα των σωματιδίων εθάλης, είναι θέμα των μειγμάτων στα οποία εκτίθεται ο κόσμος, όπως για παράδειγμα το όζον, που δεν είναι καλό για τον άνθρωπο αλλά και για τα οικοσυστήματα και για τα φυτά. Και πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, εντάσσουμε τα μέσα αυτά στην ε, μελέτη αντικτύπου. Να λάβουμε υπόψη περισσότερα ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τόπων, όχι να αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη ως ένα σύνολο. Θα πρέπει να είμαστε πιο... να λαμβάνουμε υπόψη μας τις διάφορες αστικές περιοχές και αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη σε ό,τι αφορά την έκθεση και τα στατιστικά στοιχεία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τις αστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και με ενθαρρύνει το γεγονός ότι η Eurostat συμφώνησε να προβεί σε στατιστικά στοιχεία βάση τόπου για να δούμε στο επίπεδο κάτω από το επίπεδο υποχρεωτικής αναφοράς των στοιχείων, τι γίνεται στο εσωτερικό των πόλεων, ακόμα και σε μικρότερους δήμους, για να έχουμε πολύ καλύτερη κατανόηση του τι σημαίνει μόλυνση στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Νομίζω ότι αυτά θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο επόμενο έτος και νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν μιλάτε για το πώς θα προσεγγίσουμε το κοινό, τον κόσμο. Πρόθεσή μας είναι να πάμε πέρα από την, ε, τις συνηθισμένες υποχρεώσεις ε, αναφοράς και να διαθέσουμε τις πληροφορίες αυτές με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Έχουμε την ε, δημόσια υπηρεσία Ion Earth που θα διαθέσει λοιπόν αυτές τις πληροφορίες στα τηλέφωνα, στα, στους υπολογιστές προκειμένου ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή και να βλέπει σε τι εκτίθεται. επίσημη. Επίσης, σε ό,τι αφορά την, ε, τον εξυγχρονισμό ενός πολύ γραφειοκρατικού συστήματος αναφοράς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχει και το κοινό σε ό,τι αφορά την υποχρέωση αναφοράς. Αυτό τι σημαίνει ότι θα διαθέσουμε φθηνού αισθητήρε μέσω τηλεφώνου, μέσω άλλων συσκευών, προκειμένου να ενημερωνόμαστε για την κατάσταση σε κάθε τόπο. Και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να, συμμετάσχουν, να συμμετέχουν και αυτοί στην διαδικασία αναφοράς των φαινομένων ως προς το περιβάλλον. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή του κοινού και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι δυτή αυτή η προσέγγιση και να είναι διτός αυτός ο διάλογος, να έχει να ακούμε και να δίνουμε πληροφορίες. Χαίρομαι που οι συναδελφοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούνται πολύ με θέματα βιοπικιλότητας και κατά πάσα πιθανότητα στην ε, πρόταση θα συμπεριληφθούν τέτοια ζητήματα. Ο κόσμος ε, θα έχει δυνατότητα να καταγράφει και να παρατηρεί ξένα είδη για να ε, καταγράφονται οι αλλαγές. Για να περάσω τώρα στη συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος, αλλά και τα θέματα βιοκαυσίμων και του καθεξής. Για να απαντήσω στην ερώτηση που θέσατε κύριε Ντέιβις για την Ιταλία. Ναι, είναι στον κατάλογο στην τελευταία έκθεση. Δεν θα ήθελα να πω ότι όλα είναι βίωνα. Αντιθέτως, γίνονται όμως βασικές αλλαγές στη δομή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ενεργειακή κατανάλωση και υπάρχει μια μετατόπιση προς το αέριο και όντως οι εκπομπές σχεδόν αποκλειστικά στην ενέργεια οφείλονται, αλλά η οικονομική δραστηριότητα κατά τα φαινόμενα είναι 2,4% αλλά έχετε δίκιο πέρα από αυτό κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε στο 25%. Η ανάλυση μας η σημερινή λέει πως ναι, μπορούμε να υπερβούμε το στόχο του 20%. Ότι είμαστε σε θέση να πετύχουμε το στόχο του 25%. Αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο προαπαιτεί συνεχιζόμενη πίεση στα κράτη-μέλη και το βλέπουμε κάθε χρόνο ότι πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αλλά για τις προτάσεις, την ομοθεσία και τον τρόπο που εφαρμόζονται τα κίνητρα, αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, θεωρούμε ότι το 25% αποτελεί ένα επιτεύξιμο στόχο και αυτό δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Υπάρχει και μια λεπτομερής ανάλυση στην έκθεση και ευχαρίστως να σας παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά και πόσο αξιόπιστα είναι. Και αυτά εντάσσονται σε ένα μοντέλο που έχει συμπεριλάβει και κάποιους παράγοντες αβεβαιότητας. Θεωρούμε μέχρι το 2020 είναι, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτό σε ώρα σε ό,τι αφορά το σύστημα ανταλλαγής ρήπων. Θεωρούμε ότι στην επόμενη φάση, σε ό,τι αφορά την κατανομή των ε, προσπαθειών, θα πετύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη γεωργία, έχω υπόψη μου και τη συζήτηση η οποία διεξήχθη. Έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στην γεωργία σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Αυτό φυσικά πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά έχει να κάνει φυσικά και με την τιμή των ε, λιπασμάτων. Άλλα θέματα αφορούν το νερό και την βιοπικιλότητα. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα μετά από πολλά χρόνια ότι γίνονται προσπάθειες και σε άλλους τομείς της πολιτικής. Οι προσπάθειες λοιπόν των τελευταίων χρόνων ε, μοιραία έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε άλλους τομείς ε, υπάρχουν θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και νομίζω ότι ως Επιτροπή και εμείς από πλευράς μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να το τονίζουμε αυτό για να μην χαθεί αυτή, αν θέλετε, η σύνδεση και με άλλους τομείς της πολιτικής σε ό,τι αφορά τα ύδατα, το νερό. Η ποιότητα των υδάτων αποτελεί, εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε ασωτούχα, έχουμε άλλα ζητήματα πολλά, αλλά διαπιστώνουμε επίσης ότι στον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων η αποδοτικότητα στη χρήση του νερού θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού. Άρα θεωρούμε ότι θα βοηθηθούμε γιατί με τη σωστή άρδρευση, αν σκεφτείτε πόσο καταναλώνεται, πόσο, από ποσοστό του νερού καταναλώνεται στην άρδρευση, 80% στο νότο, πολύ απλά ε, θα πρέπει να προσέξουμε πόσο νερό διαθέτουμε στο σύστημα και φυσικά και πολλοί αγρότες εξετάζουν τις άλλες ε, δυνατότητες που έχουν λόγω της υψηλής συγκέντρωσης. Και άρα θεωρούμε ότι το συνολικό φόρτος θα περιοριστεί και έχουμε ήδη κάποιες τέτοιες ενδείξεις στις νότιες χώρες. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα της ε, βιοπικιλότητας και γενικότερα πώς μπορούμε να θέσουμε πολιτικές ε, που μπορούν να πετύχουν. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι το εξή. Η βιοπικιλότητα έχει και το κόστος της ε, ανάκτησης του πληθυσμού. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο θεωρούμε ότι δεν ε, αξιοποιείται επαρκώς σε ό,τι αφορά την ανάλυση αντικτύπου. Και γιατί το αναφέρω, γιατί το κόστος αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του λογιστικού συστήματος των οικοσυστημάτων, αν θέλετε. Και έτσι γίνεται η σύνδεση με το σύστημα των εθνικών λογαριασμών. Με ένα... με μία σειρά μετατροπών μέσα στυλών μέσω ένας, με ενός κόστους ανάκτησης. Και αν το κόστος αυτό, μάλλον αν θέλουμε να προχωρήσουμε και ελπίζω το Κοινοβούλιο να δει και να διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα της λογιστικής αυτής, νομίζω ότι μόλις ενταχθεί αυτό το κόστος ανάκτησης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν επιχειρήματα κατά της βιοπικιλότητας. Να μην ληφθεί υπόψη, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την πράσινη, ε, τις πράσινες υποδομές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να τονίσουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις πολιτικές αυτές και για την βιοπικιλότητα και για τον αέρα και για το νερό. Τώρα, για τα βιοκαύσιμα, τη βιοπικιλότητα, τη βιομάζα και την... Ε, είναι σαφές ότι όταν επισερχόμαστε σε προς ε, συζητήσεις για τα βιοκαύσιμα και κατά πόσον είναι ουδέτερα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, καταλήγουμε στο εξής καταλήγουμε σε βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση αναφοράς. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω όταν με ρωτούν κατά πόσο μπορούμε να καταρτήσουμε κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα είναι ότι ναι, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει ε, αποκαλύπτοντας πλήρως τι καλλιέργειες γίνονται και αυτό περιλαμβάνει και πλήρη συμμετοχή των χωρών. Δεν είμαι βέβαια ότι σε πολιτικό επίπεδο ρημότητας είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και δεν θα μπορούσα να σας πω ότι στην παρούσα φάση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δορυφορικές εικόνες ή κάποιες εκτιμήσεις για να σας δώσω τη βεβαιότητα την οποία θα χρειαζόσασταν για να, θέσετε τα κριτήρια που χρειάζεστε. Και αυτό αποτελεί ένα δίλημα ειλικρινά για μένα. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Ε, τι χρειαζόμαστε για να συζητήσουμε με κάθε χώρα πώς παράγει τη βιομάζα που παράγει. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετική συζήτηση και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε τη χρήση των γεών και πώς μπορεί να αλλάξει αυτή εν μέρη, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση ε, σε ό,τι αφορά τις πράσινες υποδομές και πώς μπορεί να αλλάξει η χρήση των γεών, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, ΚΑΠ. Μπορεί να ενέχονται κίνδυνοι στο να πούμε ότι, για παράδειγμα, θα κρατήσουμε την ε, χυψή καλλιέργεια το θέμα λοιπόν είναι το πώς θα προδιαγράψουμε αυτή τη βιωσιμότητα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά όμως τις διεθνείς συζητήσεις που ενδιαφέρει τους πιο πολλούς από εσάς, θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη πολιτική βούληση, βούληση προτού μπορούμε να πούμε ότι η βιομάζα πραγματικά είναι ουδέτερη. Και να περάσω στο πρακτικό ζήτημα τώρα των αποβλήτων και του ρόλου του οργανισμού. Ξέρω ότι μιλήσατε για, το, για την υπηρεσία εφαρμογής ζητημάτων αποβλήτων. Το θέμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή είναι ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Φυσικά υπάρχει ένα πολύ βασικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την μη μεταφορά από νομικής άποψης. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να παίξει το ρόλο της για να καλέσει σε συζητήσεις τα κρατημέλη αλλά θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα με τα απόβλητα, γιατί έχω μεταβεί σε πολλέ χώρε πλέον και έχω εξετάσει τα θέματα εφαρμογή της νομοθεσίας των αποβλήτων, είναι ότι υπάρχουν επτά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν επιτάπητο. Η μη συμβατότητα, η έλλειψη επενδύσεων, η έλλειψη ικανοτήτων σε πολλές περιπτώσεις κυριολεκτικά, οι παρανοήσεις που επικρατούν για τα βασικά, τις βασικές αρχές μεταξύ της ανακύκλωσης, της εκ νέου χρήσης κτλ. Είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακό πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των φιλοδοξιών που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και της πράξης. Επίσης, υπάρχει μεγάλη παρανόηση για το τι, ε, πώς θα πρέπει να κατατάσσονται τα απόβλητα ανά χώρα, ε, δεδομένου και του πληθυσμού, δεδομένου και των ιδιωτήτων της κάθε χώρας. Άρα, αυτό που θα πρότεινα είναι την επόμενη περίοδο, την επόμενα ένα-δύο έτη ίσως, νομίζω ότι καλύτερο να κάνουμε κάποιες πιλωτικές έρευνες, εξετάζοντας την πλήρη έκταση και την ακριβή έκταση του προβλήματος, γιατί έχοντας μεταβεί στις χώρες που έχω πάει, διαπιστώνω ότι πολλά θέματα εφαρμογής θα μπορούσαν να επιληθούν με πολύ άμεσο και πρακτικό τρόπο, χωρίς τεράστιο, ε, τεράστια προσπάθεια, αν θέλετε, χειραγώγησης. Και νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να συζητήσουμε με τις χώρες και να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα εφαρμογής. Αυτό θα ήταν πιο πρακτικό παρά να επιβάλλουμε μια επιπλέον ε, ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι ο έλεγχος. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών. για την ποιότητα τη ατμόσφαιρας νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν πιο πολύ οι δήμοι και οι κοινότητες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά για τα απόβλητα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός με, με το δίκτυο που έχει στα κράτη-μέλη. Αυτό θα απαιτήσει φυσικά πιο πολλούς πόρους, αλλά θεωρώ ότι με πολύ καλύτερη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά τους επόμενους έξι μήνες και να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο πώς ε, θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή. Νομίζω ότι κάλυψα όλους τους τομείς ε, που μου θέσατε ερωτήσεις, αλλά ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, Ζακλίνα. Ε, πραγματικά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η υπηρεσία σας και η δουλειά μας η ίδια εξαρτάται από τις μελέτες και τις δικές σας αναλύσεις. Και όπως βλέπετε όλες οι ερωτήσεις ετέθησαν ποιότητα της ατμοσφαίρας, ε, των νερών, τα απόβλητα, το επόμενο θα είναι τα προβλήματα με τις κομματερές σε διάφορα κράτη-μέλη, να δούμε πώς γίνεται η παρακολούθηση και η υλοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ενθουσιάστηκε η αντιπροσωπεία από την υποδοχή που τους επιφυλάξατε στην Κοπεχάγη. Θα συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία, καλή τύχη. Πραγματικά σας χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε την ικανότητα και ε, την εργασία του οργανισμού στην Κοπεχάγη. Θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Yes, see you next time. See you <laughs> λοιπόν, είστε επανειδήν. Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξή μας με το θέμα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον στα διάφορα Πρώτο θέμα, η κατάσταση στην Ελλάδα. Ο κ. Σκυλακάκης είναι εδώ. Ναι. Είναι εδώ. Κύριε Σκυλακάκη, έχετε το λόγο. Ορίστε. Well, my uh, is... Είναι απλό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούσε την εφαρμογή της οδηγίας 9156 για τα απόβλητα και κυρίως το κλείσιμο των εφισταμένων χιτά στην ε, Ελλάδα. Είναι μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μου. Οξύ αυτή τη στιγμή, αρκετά οξύ. Λοιπόν, οι παράνομες χωματερές έπρεπε να είχαν κλείσει τέλος Ιουνίου 2011 και προθεσμία για την ε, αποκατάστασή τους είναι Ιούνιος 2012. Η Επιτροπή είπε ότι θα αναλάβει ένα τα μέτρα και να προσφύγει ακόμα και στο δικαστήριο. Ερώτημα. Ποια είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα, πόσες χωματερές έκλεισαν μέχρι τώρα και πόσο πιθανό είναι να σταματήσουν όλες οι χωματερές μέχρι το να κατασταθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Λειτουργούν κανονικά μέχρι τον Ιούνιο του, τον του 2012. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει σε αυτό το πρώτο σημείο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λάβαμε την τελευταία έκθεση των ελληνικών αρχών στις 26 Ιουλίου και επιβεβαιώνει αυτή η έκθεση ότι οι ελληνικές αρχές ξέφυγαν από την προθεσμία για να κλείσουν τα πάντα μέχρι 30 Ιουνίου του 2011. Σύμφωνα τις αρχές εξακολουθούν να υπάρχουν 82 παράνομες χωματερές που είναι ανοιχτές από, από 361 το 2009 που ήταν 369 Μεγάλη πρόοδος, αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά και υποσχέθηκαν οι αρχές να κλείσουν τα πάντα μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Συναντηθήκαμε με τις ελληνικές αρχές στις 14 Σεπτεμβρίου, μας εξήγησαν ότι η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα της μεταρρυθμίσεως στους Δήμους. Ήταν ένα μοναδικό πρόβλημα, ενίο πρόβλημα. Έκαναν τα πάντα για να καθαρίσουν οι χωματερές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πολύ χαμή ρυθμοί απορρόφηση χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι χωματερέ, αλλά ο ρυθμό απορρόφηση είναι περίπου 6 8% αν δεν σφάλω. Γι' αυτό ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε task force για την Ελλάδα. Ένα από τα καθήκοντα τη task force ήταν να βοηθηθούν οι ελληνικέ αρχέ να χρησιμοποιήσουν γρήγορα του πόρου Ευρωπαϊκή Ενώση για να αποκατασταθούν οι χωματερέ και εξέδωσε ανακοινωθέν τύπου στις 13 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή IP 11 για την πρώτη συνάντηση μεταξύ Task Force και ελληνικών αρχών. Δύο φορές αναφέρεται, αναφέρονται, αναφέρεται η διαχείριση των αποβλήτων. Εξακολουθεί να υπάρχει η διαδικασία αυτή για παράβαση. Επόμενη διαδικασία είναι η παραπομπή στο δικαστήριο για επιβολή κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως εστιάζεται μέσω της Task Force να διατεθούν περισσότερο, να απορροφηθούν περισσότερο δυνατοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να κλείσουν οι χωματερές να, και να γίνει αποκατάσταση των περιοχών αυτών μέχρι τον τέλος Ιουνίου του 2012. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση αν είναι εδώ για το θέμα των αποβλήτων για την καμπανία, για το θέμα των αποβλήτων στην καμπανία στην Ιταλία. Υπάρχει κάποιος να τον εκπροσωπήσει. Πάμε στο ερώτημα του Chris Davis. Για τις περιοχές Natura 2000 στη Βουλγαρία, Chris, έχει το λόγο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν το περίμενα αυτό. Φτάσαμε στην ερώτηση 5 εντός 5 Βουλγαρία. Ποιος είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, ευχαριστώ. Στην Επιτροπή ετέθη το θέμα εδώ και ένα εξάμεινο περίπου και είπαμε τότε θα ζητήσουμε να επανέλθετε. Ευχαριστώ που επανήλθατε. Όταν μας δόθηκε προηγούμενη απάντηση, μου είχε εντύπωση ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επίτροπη το γνώριζε το πρόβλημα, δεν γινόταν πολλά πράγματα. Έκτοτε υπήρξε πρόοδο και ελπίζω να τη σχολιάσετε. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Καλωσορίζω την επιτεθήσα πρόοδο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βήματα που έκανε για εξασφαλίσει το ότι εφαρμόζεται σωστά ο νόμος, αλλά θα ήθελα να πω επίσης ότι από τώρα μέχρι προσφυγή ενδεχόμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει χρόνος μεγάλος και μπορούν να πάνουν πολλά στραβά με αυτή την περιοχή. Πήρατε κάποια βήματα για να ενθαρρύνετε τη βουλγαρική κυβέρνηση ούτως ώστε να προστατευτούν αυτές οι περιοχές και ανάπτυξη ε, εγκαταστάσεων αιωλικής ενέργειας να περιοριστεί, να συγκρατηθεί μέχρι ότου γίνει η σωστή αξιολόγηση. Ευχαριστώ, Κρίς, για αυτή την ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει την καλοσύνη να απαντήσει. Ευχαριστώ, ναι, πράγματι, όπως είδατε, επιτεύχθη πρόοδος από την προηγούμενη φορά. Έξι ζώνες είχαμε, όπου υπήρχε πρόβλημα καθορισμού, για τις τέσσερις έχουν καθοριστεί από τις αρχές Έχουμε δύο εκρεμή ζητήματα. Καλλιάκρα και Ρίλα. Η, η Ρίλα δεν υπάρχει προγραμματισμό για ολική ενέργεια στο Καλλιάκρα. Έγινε επίσκεψη αποστολή από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος τέλος Αυγούστου. Συλλέξαμε πληροφορίες, στοιχεία, εικόνες διαφόρων αιωλικών τουρμπινών. Θα δείτε αρκετά εντυπωσιακέ εικόνες. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπροματική ειδοποίηση τέλος Σεπτεμβρίου γιατί δεν υπήρχε αιτιολογημένη άποψη ακόμα, διότι θέλαμε νόσημα τα στοιχεία, έλλειψη καθορισμού, οικοδόμηση σε αυτές τις περιοχές τουρμπινών, ακόμα και γήπεδο γκολφ. Έχουμε λοιπόν το φάκελο, τεκμηριωμένο, θέλουμε να δούμε τι θα απαντήσουν οι αρχές μέχρι τέλος Νοεμβρίου και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε. Όπως αναφέρατε στο ερώτημά σας για την ώρα, υπάρχει ένα πάγωμα μορατόριου όσον αφορά τις ε, ολικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Είναι εν μέρη η πολιτική απόφαση του Υπουργού και εν μέρη έλλειψη δυνατότητα παραγωγής τεχνικής ενέργειας το κίνητρο για την κατασκευή αυτών των μονάδων παραγωγής ηλικής ενεργείας. το δίκτυο δεν θα σηκώσει παραπάνω τουρμπίνε ολική ενέργεια, οπότε εκεί είμαστε ασφαλεί για την ώρα. Θα δούμε, όπω σα είπα, τι θα γίνει αργότερα. Για, το Ρίλα, για τη Ρίλα θα αποφασιστεί η δράση την επόμενη εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντα την ίδια γραμμή. Ε, θα στείλουμε ε, σημείωμα ε, ενημερωτικό κλπ. Και, θα δούμε πώ θα κινηθούμε. Κάτι συμπληρωματικό όσον αφορά την, την κατάσταση. Εξετάζουμε και από τι δύο πλευρέ των σύνορων τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται με ολικές μονάδες και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Και ξεκινάει και διαδικασία παράβασης κατά της Ρουμανίας για το ίδιο πρόβλημα. Και έγινε, δημιουργήθηκε task force για να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των μελών. και τελικά να παραδείγματο χάρη ότι ως πτηνά τη γλιτώσουν από την ε, Βουλγαρία, από την Ατούρα να μην περάσουν και συλληφθούν από τις τουρμπίνες στη ε, Ρουμανία. Ε, δύσκολο να καλύψει κανείς την ύπαρξη αιωλικής εγκατάστασης ή πολλών αιωλικών τέτοιων μονάδων. Γι' αυτό μπορέσατε να μαζέψετε στοιχεία που θα είναι πιστικά αν τελικά υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο, γίνει προσφυγή. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, υποθέτω. Ποτέ δεν πήγα σε αυτή την περιοχή, αλλά φαντάζομαι ότι αν υπήρξε ανάπτυξη ολικής ενέργειας σε σημαντικό βαθμό και κάτι που αντιβαίνει τον καθορισμό της περιοχής αυτής σαν προστατευμένη, τότε τελικά ίσως να ζητήσετε να απεγκατασταθούν αυτές οι μονάδες παραγωγής. Όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά, τα πράγματα γίνονται πολιτικά πολύ δύσκολα. Και θα με ενδιαφέρε, θα ενδιαφερθώ, θα ήθελα να ξέρω πώς θα κινηθεί όσον αφορά αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να απαντήσετε. Θα έμπαινε στον πειρασμό να πω ότι είναι υποθετικό αυτό. Αλλά εγώ θα λέγω ότι τι επιλογές είναι ανοιχτέ. Και γιατί ετοιμάζουμε και τεκμηριώνουμε την υπόθεση και συλλέγουμε στοιχεία είναι διότι θέλουμε να έχουμε δυνατότητες επιλογής εάν θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε διαδικασία αυτή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, αυτό με βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, ο κύριο Ρώση κατέφτασε, του δίνω το λόγο για την εφαρμογή τη οδηγία για τα απόβλητα στην περιοχή τη καμπάνια. Ήθελα πληροφορίες αφής όσον αφορά την πολύ πρόσφατη ε, θέση προειδοποίησης της Ιταλίας όσον αφορά τα απόβλητα στην ε, Καμπανία. Θα ήθελα να με ενημερώσετε τι γίνεται τελικά με την όλη κατάσταση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αναφέρω δύο πράγματα. Πού βρισκόμαστε αφορά τη διαδικασία για την Ιταλία Ρωτήθηκε και ποια είναι η άποψή μας, η εξολόγηση της καταστάσεως στην καμπανία διαδικαστικά. Όπως τα παρατήρησε το αξιότιμο μέλος, έστειλε μία επιστολή του άθου 260, δηλαδή με άλλα λόγια επόμενο βήμα θα είναι έτοιμα προσφυγής στο δικαστήριο με έτοιμα επιβολής οικονομικών κυρώσεων. Πού βρισκόμαστε η Ιταλική κυβέρνηση έστειλε διαχειριστικό σχέδιο την περιοχή Καμπανίας. Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Καμπανίας τέλος Μαρτίου. Αναδημοσιεύθηκε μέσα Ιουνίου. Σχέδιο κειμένο όμως. Όμως δεν τίποτα παραπάνω. Γίνεται περιβαλλοντική στρατηγική ανάλυση και τελικά στο κείμενο υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Λέω ότι είναι σχέδιο κειμένου γιατί δεν έχει οθετηθεί ακόμα. Και δεύτερον, όσον δεν εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο, μπλοκάρονται τα χρήματα που πηγαίνουν για ενίσχυση της καμπανίας. Αυτό θέλει η τελική κυβέρνηση. Πώς αξιολογούμε εμείς την κατάσταση. Στείλαμε λοιπόν αυτή την επιστολή του άρθρου 260 που σημαίνει ότι, ότι δεν μας ικανοποιεί το σχέδιο διαχείρισης ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση τελικά θα, θα επικρατήσει το κοινοτικό δίκαιο αν εφαρμοστεί το σχέδιο διαχείρισης, εάν εφαρμοστεί. Δεν φτάσαμε όμως εκεί ακόμα. Το πρόβλημα με τις χωματερές είναι να σταματήσει η παραγωγή των αποβλήτων η συλλογή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό δεν έχει γίνει ο διαχωρισμός των αποβλήτων, ο, ο ρυθμός συλλογής διαχωρισμένων αποβλήτων είναι πολύ ε, μικρός όσον αφορά αναρεοβικά συστήματα χωνευτήρια στο Σαλέρνο υπάρχει μόνο ε, μία τέτοια μονάδα, εννιά άλλες πρέπει υποτίθεται να κατασκευαστούν, δεν έχουν κατασκευαστεί, καυστήρες στη Καζέρτα, Σαλέρνο και στην Νάπολη υποτίθεται ότι το 2014 θα ε, αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι μονάδες αποτέφρωσης αόριστη η χωρητικότητα των χωματερών που υπάρχει μέχρι τώρα και έχουμε 6 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων που έχουν σωσαρευτεί. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τεφρωτής, από τεφρωτήρας. 2014 λέει η κυβέρνηση. Πρόβλημα. Έλλειψη λύσεων όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο 7.200 τόνοι καθημερινά αποβλήτων παράγονται στην καμπανία. Στη, από τις υψηλότερες παραγωγές αποβλήτων στην Ιταλία. Συνεργαζόμαστε Ιταλικές αρχές σε όλα τα επίπεδα. Ο Επίτροπός μου συναντάται τακτικά με τις αρχές. Προσπαθούμε να πιέσουμε τις Ιταλικές αρχές προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η κατάσταση. Όταν εθετηθεί το σχέδιο διαχείρισης θα έχουμε πρόοδο, εν τω μεταξύ κινδυνεύουμε να δούμε εικόνες από το παρελθόν, από σκουπίδια στους δρόμους. Ελπίζουμε η δίκηση να το αποφύγει αυτό, η κυβέρνηση, αλλά ακόμα υπάρχει αυτή η διαδικασία παράβαση και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Κάντενμπαχ, δύο ερωτήσει έχετε αν δεν απατώμε για την Natura 2000. Στα αγγλικά. Μάλιστα, να αρχίσω από τη διαφάνεια. Η Αυστρία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει δώσει στοιχεία ε, για την Natura 2000 ε, ούτε στο viewer ούτε στη βάση δεδομένων. Κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό συνιστά παραβίαση της ε, οδηγίας 2003 4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. Είναι η ερώτηση παριθμών 3 της κυρίας Κάντενμπαχ. Θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ κύριε. Μπορεί να ε, παραβιάζει το πνεύμα, αν μη τι άλλο, τις οδηγίες για τη διαφάνεια. Γνωρίζετε ότι δύο κράτη-μέλη αντιτίθενται στη δημοσίευση αυτής της πληροφόρησης για την Natura 2000. Το άλλο κράτος ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει αποσύρει τώρα την αντίσταση. Και η Αυστρία είναι η μελανή κοιλίδα, ε, αν θέλετε, τροποτίνα. Το έχουμε θέσει υπόψη των Αυστριακών Αρχών τέλη Σεπτεμβρίου και μας υποσχέθηκαν να κάνουν κάτι. Κατά την άποψή μου, ε, μάλλον εξ όσων γνωρίζω, ε, διαφωνούν ένα ή δύο κρατήρια. κρατήδια. Και επειδή ε, είναι τέτοιο το σύστημα λήψη αποφάσεων στην Αυστρία, αυτά τα δύο κρατήδια μπορούν να μπλοκάρουν το σύνολο της απάντησης. Για την ε, οδηγία λοιπόν περί διαφάνειας 2003 4 υπάρχει ένα άρθρο 7 εδάφιο 2β που ε, ομιλεί για ευρία διάδοση των σχεδίων και των προγραμμάτων. Ε, από απονομική απόψεως δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο και αν παραβιάζεται το γράμμα της οδηγίας, αλλά ζητούμε από τις αυστριακές αρχές να δημοσιεύσουν τα στοιχεία αυτά. Εξακολουθούμε να πιέζουμε και από πλευράς ε, πολιτικής και το πνεύμα του άρχους, αλλά και από νομικής πλευράς βλέπουμε το θέμα αυτό της οδηγίας περί διαφάνειας. Όπως γνωρίζετε, η Επίτροπός μου ενδιαφέρεται πολύ ε, για το θέμα του περιβάλλοντος. Και καλό είναι η Αυστρία να λύσει αυτό το πρόβλημα το συντομότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία μπαχ. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στην επόμενη ερώτηση. Η εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 στην Αυστρία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Σύμφωνα με την ενημερωμένη λίστα αποθεμάτων και ε, οικοτόπων για τα είδη, παραμένει ο ε, ορισμός ε, πέντε <clears throat> οικοτόπων στις Άλπεις και 12 αλλού στην Αυστρία η διαδικασία προσφυγής κατά της Αυστρίας της 11 η του 2008 το Δεκέμβριο του 2009 αποσύρθηκε λόγω ελλείψεως αποδεικτικών στοιχείων. Πότε θα ξαναρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δράση της κατά ε, της ε, Αυστρίας. Κοιτάξτε, απάντηση. Ε, η δουλειά θα πρέπει να γίνει ε, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της επιβολής ε, του περιβαλλοντικού δικαίου είναι ότι συνδέεται με επιστημονικά στοιχεία. Όταν ε, αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία κατά της Αυστρίας, θεωρούσαμε ότι είχαμε επιστημονικά στοιχεία και διαπιστώσαμε ερχόμενοι ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν υπήρχαν. Ξέρουμε ότι πάει στραβά εκεί, γιατί... Ε, είναι υψηλότερο το επίπεδο μη ορισμού αυτών των, ε, ή χαρακτηρισμού αυτών των περιοχών στην Αυστρία σε σχέση με άλλες χώρες ε, σε ό,τι αφορά τις ρεζέρβες ας πούμε και τις προστατευόμενες περιοχές και οικοτόπους αλλά θα πρέπει να ε, οριστούν σαφώς ξανά αυτές οι περιοχές και το μελετούμε πολύ προσεκτικά πριν προσφύγουμε στο δικαστήριο γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε. Γι' αυτό αποσύραμε την υπόθεση. Δεν θέλουμε να τη χάσουμε προφανώς το ΔΕΚ και έχουμε ακόμα τη δυνατότητα τώρα, έχοντας αποσύρει αυτή τη διαδικασία, να επανέλθουμε όταν θα έχουμε αδειάσει τα στοιχεία. Η δυσκολία ποια είναι. Ότι το δικαστήριο είναι πολύ πιο αυστηρό απέναντί μας. Πέρυσι, ε, σε σχέση με τον Ισπανικό Λίγκα, ε, αντιμετωπίσαμε ε, μεγάλα προβλήματα στο δικαστήριο, ε, είναι πολύ αυστηρή μαζί μας, δεν θέλουμε να ξαναρχίσει αυτή η κατάσταση του χρόνου. Γιατί δεν προχωρεί το συγκεκριμένο θέμα, γιατί εμείς από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να έχουμε αδιάστα, όπως σας είπα, επιστημονικά στοιχεία για να μπορούμε να τα τεκμηρώσουμε στο δικαστήριο. Κανένα χρονοδιάγραμμα μπορεί να μας δώσετε, λέει κυρία Κάντεμπαχ, όχι απλώς του χρόνου. Ε, αυτό θα το ρωτώ και ε, από τους συναδέλφους που χειρίζονται το θέμα το πρώτο εξάμεινο του 2012 πιο συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω πρέπει να στοιχειοθετήσουμε πολύ τα ε, στοιχεία αυτά ε, ανάλογα με το είδος το είδος και οικότοπο προς οικότοπο υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνετε το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα την Επιτροπή μας και να μην χρειάζεται κάθε εξάμεινο να σας κάνουμε τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. λοιπόν, νομίζω ότι Τελειώσαμε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν το 6 και προτείνω να περάσουμε στο επόμενο. Περιορισμό των εκπομπών πτυτικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει το κείμενο. Ο κύριος ε, Τόμας Φερέιε, αν θέλετε να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ, περί πρόκειται. Yes, good afternoon. Καλησπέρα σας. Εγώ εκπροσωπώ τον Τόμας Περχέιε και λέγομαι Φιλίπ Φρανσουά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσετε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας 2004 42 ε, που είναι καλύτερα γνωστή ως οδηγία χρωμάτων, η Deco Paints, 25 Μαΐου ε, εγκρίθηκε. Θα ήθελα να θυμίσω λίγο το ιστορικό της οδηγίας αυτής. Η οδηγία για τα χρώματα έχει στόχο να περιορίσει τις εκπομπές πτυτικών οργανικών ενώσεων. VOC λέγεται αυτό στα αγγλικά, γιατί έχουν οργανικούς διαλύτες και είναι ε, σε χρώματα διακόσμησης, βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων. Αυτές οι πτυτικές οργανικές ενώσεις ε, στον αέρα δημιουργούν ε, επικίνδυνα φωτοχημικά παράγωγα, όπως είναι το όζον στη στρατόσφαιρα. Ε, λόγω λοιπόν αυτής της ρήπασης υπάρχει οδηγία για ε, τα οριακές τιμές ανώτατες των εκπομπών που από το 2010 και μετά θα πρέπει να τηρούνται και αφορούν τις πτυτικές οργανικές ενώσεις, τα VOCs. Τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορες πηγές λοιπόν εκπομπών και αυτά είναι και προϊόντα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν αυτά τα μέτρα στα, σε επίπεδο κρατών μελών και εμεί ερχόμαστε να τα συμπληρώσουμε. Η θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρήπαση του 2005 θεώρησε ότι θα πρέπει να μειωθεί κατά 51% η οριακή τιμή σε σχέση με τα επίπεδα του 2000 για να φτάσουμε στους ενδιάμεσους στόχους του 2020 που έχουν ε, οριστεί στην παρούσα θεματική στρατηγική. Η ευρύτατη λοιπόν εκτίμηση θεώρησε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί το υφιστάμενο και εκτιμένο και αυτή η οδηγία περί χρωμάτων έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Ζητεί λοιπόν η οδηγία αυτή τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή να ε, μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά όταν οι φυτικέ οργανικέ ενώσει ε, δεν υπερβαίνουν μία οροφή. Από την 1η Ιανουαρίου του 2007 ισχύει αυτό. Για τι βαφέ και τα βερνίκια από την 1η Ιανουαρίου 2010 είναι πιο αυστηρές ακόμα οι τιμές. Η οδηγία επίσης ε, επιβάλλει την επισήμανση ε, των προϊόντων αυτών. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της, οι πρώτες εκθέσεις από τα κράτη-μέλη για τη διαδικασία παρακολούθησης πρόκειται να κατατεθούν τον Ιούνιο του 2008 και αφορούσαν το έτος 2007. Τότε ε, η υλοποίηση της οδηγίας ήταν ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο και τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν προσωρινά και πρόωρα. Οι εκθέσει των κρατών μελών μα έδωσαν στοιχεία ότι τα κράτη-μέλη παρακολουθούν την εφαρμογή με επιτόπιε ε, δειγματοληψίες, επιθεωρήσεις και ελέγχους. Ωστόσο το 2007 κάποια κράτη καθυστερούσαν ε, στην υλοποίηση προγραμμάτων επιθεώρησης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> τους ενθάρρυνε να ε, μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Περαιτέρω πληροφόρηση θα συλλεγεί από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή το 2010 ε, οι εκθέσει που κανονικά έπρεπε να κατατεθούν μέχρι το θέρο. Θα τι αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τις συνοψίσει στην επόμενη έκθεσή μας που αναμένεται στα μέσα του 2012. Το άρθρο 9 της οδηγίας ζητάει αυτή την αναθεώρηση για να δούμε κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η εκπομπή αυτών των ε, οργανικών ε, ουσιών. Το 2008 και 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> έκανε μια μελέτη που καλούσε όλους τους ενεχομένους να ε, μελετήσουν όλα τα ενδεχόμενα ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και να υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια για την οριακή τιμή σε ό,τι αφορά τα προϊόντα φωνοποίησης αυτοκινήτων. Οι περιορισμοί στις εκπομπές ήταν μικρή, ενώ το γραφειοκρατικό κόστος και άχθος ε, ιδιαίτερα αυξημένο. Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η αναθεώρηση ε, του πεδίου εφαρμογή ή των οριακών τιμών αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται. Αυτό είναι ένα προκατακτικό συμπέρασμα το οποίο θα αναθεωρηθεί το 2013 όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της θεματικής στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κοιτάξει τότε τους ενδιάμεσους στόχους και για το περιβάλλον ε, και ε, κατά πόσο θα είναι σκόπιμο να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ατμοσφαιρική ρήπανση ε, και πάντα έχοντας υπόψη μας το κόστος και τη σχέση κόστους και ωφέλειας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Οκονή έχει ζητήσει το λόγο. Όχι, για το επόμενο θέμα. Άλλος? Ο κύριος Τζανώνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα την έκθεση. Είδα κάποια σημεία και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις, παρακαλώ. Όσον αφορά, λοιπόν, τους ελέγχους των κρατών μελών, τους εσωτερικούς ελέγχους, έγιναν επιθεώρηση παραγωγών εισαγωγών χονδρεμπόρων, εισαγωγέων χονδρεμπόρων, λιανοπολιτών από, από, από ελάχιστο 0 μέχρι 540 ελέγχους. Μεγάλη διαφορά ελέγχων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Που πιστεύω ότι είναι μεγάλο εμπόδιο, υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για την εφαρμογή της και πιστεύω ότι δυστυχώς είναι κοινό πρόβλημα που αφορούν και πολλές άλλες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ενδιαφέρον, πιστεύω, να σκεφτούμε ένα ομοιόμορφο σύστημα όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους, βλέποντας τις πολύ μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Στην έκθεση δεν βρήκα πίνακα στον οποίο να παρατίθεται αυτή η έλεγχη από πλευράς μελών κατά χώρα. Εάν υπήρχε ένας κατάλογος, ένας πίνακας θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον, πολύ πιο άμεσο να δει κανείς ποιος έκανε τους ελέγχους και ποιος δεν τους έκανε. Μετά διαβάζω ότι η βασική δυσκολία για την εφαρμογή της οδηγίας αφορά την έλλειψη πόρων διοικητικών που θα διατίθεται σε αυτή την δραστηριότητα της εποπτείας του ελέγχου. Διερωτώ με, έναντι μιας τέτοιας οδηγίας μήπως θα έπρεπε να προβλέπονται και κάποια ε, χρήματα ως ενίσχυση για τα κάτι μελη διότι δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι, οι οδηγίες σε καποια κάτι κράτη-μέλη δεν εφαρμόζονται. Άλλο ερώτημα, σε άλλο σημείο, Στην έκθεσή σας βλέπω ότι μια σημαντική μείωση των πτυτικών οργανικών ενός, των COVs, θα ήταν δυνατή εξαλείφοντας τα προϊόντα που υπάρχουν στα αποσμητικά και τα αντιδροτικά. Και είπατε ότι δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, διότι δεν θα πετυχαίναμε τη συνένεση των καταναλωτών για κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι έναντι του προβλήματος της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και της υγείας θα ήταν καλό να ξεπεράσουμε αυτήν την ανάγκη για συνένεση των καταναλωτών. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχαμε συνηθίσει όλοι να χρησιμοποιούν ε, το νάιλον και, τα πλαστικ, και πλαστικές σακούλες για να κάνουν τις αγορές και αλλάξαμε τον τρόπο ζωής και δεν συνέβη τίποτα. Αντίθετα, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί να σταματήσουμε σε αυτή την περίπτωση έναντι αυτού του προβλήματος, κατά την άποψή μου, δεν είναι πραγματικό πρόβλημα. Όσον αφορά μετά τις βελτιώσεις των ελέγχων, που θεωρείτε κάτι αναγκαίο, τι έχετε πρόθεση να κάνετε. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα της εκθέσεως είναι αρκετά αδύναμα. Θα έλεγα υπάρχει σχεδόν μια παρέτηση. Εγώ περίμενα κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Όχι. Όποτε δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει απάντηση. Thank um, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα θέματα εφαρμογή και τις διαφορές στον αριθμό των ελέγχων και των επιθεωρήσεων για τη συμμόρφωση. Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια πρώτη αποτύπωση φωτογραφική, αν θέλετε, της κατάστασης. Το 2007 μας ενημέρωσαν τα κράτη-μέλη. Θυμίζω ότι η οδηγία εγκρίθηκε το 2004 και ετέθη σε ισχύ μόλις το 2007. Διαπιστώσαμε αυτή τη διαφορά ε, και την αναντιστοιχία και συστήσαμε ακριβώς ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και έλεγχο συμμόρφωσης μεταξύ των κρατών μελών για να ε, είμαστε βέβαιοι ότι γίνονται οι απαραίτητοι και σωστά έλεγχοι. Αλλά δεν θα πρέπει να προτρέχουμε σε συμπεράσματα που μπορεί να είναι πολύ νωρί από την πρώτη έκθεση. Προσπαθούμε τώρα να εκτιμήσουμε την κατάσταση σε σχέση με την περίπτωση του 2010. Να δούμε και να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για την κατάσταση εφαρμογής και σε αυτό το θέμα. Επίσης, υπάρχει και πρόβλημα διοικητικής υποστήριξης λόγω των πόρων ε, και αυτό θα το κοιτάξουμε ε, σύμφωνα με την ενημέρωση που θα μας δώσουν τα κράτη φέτος. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση και το ενδεχόμενο διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, Υπάρχει δυνατότητα σε προϊόντα φωνοποίησης για μεγαλύτερη μείωση πτυτικών οργανικών ενώσεων, υπάρχει μια υποκείμενη μελέτη που έγινε, αλλά ε, υπήρξε η αίσθηση ότι δεν έχουμε αρκετή ενημέρωση για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Δηλαδή, εάν απαγορεύσουμε αυτά τα προϊόντα, μπορεί οι καταναλωτές να στραφούν σε κάποια άλλα που να περιέχουν περισσότερες πτυτικές οργανικές ενώσεις ε, χειρότερες. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν εκεί, έλλειμμα ε, στην ε, ενημέρωση για την ε, καταναλωτική συμπεριφορά. Και θα σήμαινε απαγόρευση ή περιορισμό των ουσιών αυτών για τις συγκεκριμένες βαφές ή τα προϊόντα. Επίσης θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρήπανση και τη νομοθεσία που την αφορά θα πρέπει να τη δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο για το πώς μπορούμε να λάβουμε μέτρα όμως ε, οικονομικά για να μειωθεί αυτή η κατάσταση και η περιεκτικότητα στις φλαβερές ουσίες. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα που είναι μια πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων οι οποίοι αποσιάζουν και συνοψίζω ε, περτίνως πρόκειται. Είχαμε πρόσφατα προβλήματα, όπως γνωρίζετε, με την εσερίχια κόλλη. Το κολοβακτηρίδιο που βρήκαμε σε διάφορα τρόφιμα και αυτό έδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες στα συστήματά μας. Και η ερώτηση ήταν ε, τι διδάγματα εξάγεται από αυτά τα συμβάντα και ενδεχομένως ποιες είναι οι προθέσεις σας για το μέλλον. Euh, και πώς μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις ε, διευκρινήσεις και για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει έρθει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί φτάσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριο Βαντάικ, ο κύριο Ράιαν, κάποιο θα μπορούσε να μα ενημερώσει μέχρι να φτάσει ο συνάδελφό του. Η συνάδελφό μου, κυρία Οκονή, είχε ερώτηση. Αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι, βεβαίω θα του δώσουμε το λόγο. Ο κύριο Ράιαν ή ο κύριο Βαντάικ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα απαντήσουν. Ευχαριστώ, Τζον από ε, υπηρεσία της DG Sanko είμαι και θα ήθελα να πω ότι από πλευράς δημόσιας υγείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει τα σημαντικά διδάγματα που θα πρέπει να εξάγουμε από το περιστατικό με το E. coli. Ιδιαίτερα επειδή προετοιμάζουμε νομοθετική πρόταση για φέτος για την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για ασθένειες. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, έχει γίνει ε, με μελέτη αντικτύπου και τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης νομοθετικής πρότασης που θα εγκρίνει κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί της αρχής, αυτή η νομοθετική πρόταση θα λάβει υπόψη τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη ε, Νόσων που δημιουργήθηκε το 2004 μετά την νομοθεσία για τις μεταδοτικές ασθένειες που εγκρίθηκε το 1998. Άρα, η πρώτη βασική αλλαγή στην νομοθεσία θα είναι μια ενημέρωση για να ληφθεί υπόψη η δημιουργία ή η ίδρυση του οργανισμού αυτού. Κατά δεύτερον, θα λάβουμε υπόψη του διεθνείς ε, κανονισμούς για την υγεία. Πρόκειται για μια διεθνή σύμβαση την οποία ενέκρινε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ε, τέθηκε σε εφαρμογή το 2005. Κάθε κράτος μέλος αποτελεί ξεχωριστά συμβαλλομένο μέρος της σύμβασης αυτής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εντάξουμε τους κανονισμούς αυτούς στο κοινωτικό δίκαιο μέσω της ενημέρωσης της νομοθεσίας μας. Κατά τρίτον, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτά που συνέβησαν με την ΙΤΑ 1 1 το 2009 με την πανδημία της γρήπης. Έχουμε, κάνουμε δύο εξωτερικές ε, αξιολογήσεις το 2009 για να μάθουμε από την κρίση τότε, το 2009 και τέλος θέλουμε να εντάξουμε και τα συμπεράσματα από την κρίση η κόλαη στις αρχές του έτους. Τι άλλο προγραμματίζουμε να κάνουμε, να διοργανώσουμε ένα συνέδριο από κοινού με τις ε, αρχές ε, ε, ασφάλειας των τροφίμων το 2011 για να εντοπίσουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ε, συγκρατήσουμε από την κρίση του E. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους της ΕΦΣΑ θα καλέσουμε και τους συναδέλφους της ΕΦΣΑ και του ΕΚΠΕΝ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη των Νόσων, για να λάβουμε υπόψη όλε αυτέ τι διαστάσει και αυτά θα ενσωματωθούν στην νομοθετική πρόταση, την οποία θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τα τέλη του έτους και ελπίζουμε ότι η ενίσχυση της νομοθεσίας για τις μεταδοτικέ ασθένειες θα οδηγήσει σε μια καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα καταρχάς, την ετοιμότητα για ενδεχόμενε ε, λοιπές απειλές μεταδοτικών ασθενειών Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τον έλεγχο, την εποπτεία, σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τις μεταβατικές ασθένειες, σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη διαχείριση κινδύνων μέσω της Επιτροπής ε, της Σχετικής και τέλος, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού σε περιπτώσεις που ξεσπούν κρίσεις μεταβλητικών ασθενειών. Άρα, θα πρέπει να μάθουμε από την κρίση και του ιτα 1 και του ΙΚΟΛΑΙ e. Να λεφτεί υπόψη η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νόσων. Να ενισχυθεί η θέση μας σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την κοινή αγορά εμβολίων θα ληφθεί και αυτό το στοιχείο υπόψη στην ε, νέα νομοθεσία. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση, την ε, ενημέρωση της νομοθεσίας για τις μεταβατικές ασθένειες, την οποία την προγραμματίζουμε, προγραμματίζουμε πριν τα τέλη του έτους. Και τώρα να δώσω το λάβω στον συνάδελφό μου, τον κύριο Μίκο, που μόλις κατέφτασε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και λυπάμαι που μου άργησα. Έπρεπε να έχω έρθει πολύ πιο νωρί. Σα ζητώ συγγνώμη. Και εμεί τελειώσαμε νωρίτερα. Δεν έπρεπε να έρθει εσεί. Ε. Ωραία. Να σα δώσω λοιπόν τα στοιχεία για το ξέσπασμα και να κάνω και κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την πλευρά της, της ασφάλισης των τροφίμων. Καταρχάς, κάποια στοιχεία να επαναλάβω ότι τα συνολικά θέματα ήταν 3.910 κρούσματα η κόλαη στην Ευρώπη, εκ των οποίων 782 ανέπτυξαν τα νεφρικά συμπτώματα, τα νεφρικά ζητήματα. ...46 νεκροί κυρίως στην Γερμανία. Και υπολογίζεται ότι 812 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν σε ό,τι αφορά την καταστροφή των λαχανικών κατά τις πρώτες εβδομάδες ε, της κρίσης. Επίσης ε, απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές ε, στη Ρωσία μεταξύ άλλων. 600 εκατομμύρια ευρώ απώλειες εκεί. Η Επιτροπή Οικονομικής Στήριξης συμπεριέλαβε 210 εκατομμύρια ευρώ ως πακέτο έκτακτης βοήθειας και επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ για τα αγροτικά προϊόντα πέρα από τα 75 εκατομμύρια τα οποία ε, δίνει μαζί με τα κρατημέλη για προγράμματα στήριξης για τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των υπευθύνων για διαχείριση κινδύνου και των υπευθύνων για την ασφάλεια των τροφίμων μεταξύ ΕΦΣΑ και ΕΚΠΕΝ ήταν πολύ αποδοτική. Τα απαραίτητα δίκτυα ενεργοποιήθηκαν άμεσα και έγιναν ε, καθημερινά σχεδόν συναντήσεις συντονισμού σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και δημόσιας ασφάλειας. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αντίδραση σε τέτοιες κρίσεις ιδιαίτερα μεταξύ σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες δημοσίας υγείας και ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ε, ελέγχουμε την ποιότητα των τροφίμων, συντονίζουμε δράσεις καταναλωτών και εντοπίζουμε τους παραγωγούς. εντοπίσαμε τους παραγωγούς που ήταν η πηγή του προβλήματος στη Γερμανία. Όπως ξέρετε, η ΕΦΣΑ βοηθούσε τη... το σύστημα γοργής αντίδρασης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήταν καλή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών στα κράτη-μέλη για να εντοπιστούν να εντοπιστεί η πιο πιθανή πηγή των κρουσμάτων. Όταν εντοπίστηκε η πηγή της μόλυνσης και έγινε ο σύνδεσμος ο απαραίτητος, καταστράφηκαν τα ε, λόγω λαχανικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, από τις, από, την 6 Ιουλίου, από τις 6 Ιουλίου 2011 απογορεύτηκαν εισαγωγές από την Αίγυπτο και ε, πρότεινε μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελεγχθεί η υγιεινή επιτόπου. Δεν έχει αρθεί η απαγόρευση εισαγωγής των προϊόντων αυτών, μάλλον έχει παραμείνει η απαγόρευση εισαγωγή σπόρων, όσο η Αίγυπτο δεν πληρεί του απαραίτητου όρου. Να σα ενημερώσω ότι η Επιτροπή πρότεινε στη μόνιμη Επιτροπή για την εντετροφική αλυσίδα να παραταθεί η απαγόρευση. Προβλεπόταν αρχικά μέχρι τέλη Οκτωβρίου, εμεί θέλουμε μέχρι τέλη του έτου να παραταθεί για να είμαστε σίγουροι ότι θα πληρούνται οι όροι που θέλουμε. Τώρα, για τα διδάγματα από την κρίση. Προφανώ θα πρέπει να εξαγάγουμε διδάγματα. Καταρχάς σε ό,τι αφορά την πλευρά της ανθρώπινης υγείας. Οι συζητήσει για το πώ θα βελτιωθεί περαιτέρω το σύστημα ε, της αντίδραση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητηθεί τον Νοέμβριο. Θα συναντηθούμε με του ε, προϊσταμένους, του επικεφαλεί των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τους επικεφαλείς των σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών. Έχουμε προφανώς ε, κάποια ιδέα και κάποιες ιδέες. Είναι βασικό οι εθνικές αρχές να μην βιαστούν, να μην σπεύσουν, να δώσουν πληροφορίες για υποτιθέμενες πηγές της μόλυνσης μέχρι να υπάρχουν τα παιδευτικά στοιχεία που χρειάζονται. Ωστόσο θα πρέπει σε όλες μας τις αποφάσεις να μην ε, προκαλούμε φόβο προκειμένου να διστάζουν οι ε, και να μην προβαίνουν ενδεχομένω στα μέτρα που απαιτούνται για την ε, προστασία της υγείας των πολιτών. Θα συζητηθεί με τα κρατή-μέλη ενδεχόμενος τρόπος ενίσχυσης ε, του κοινωτικού συστήματος σε ό,τι αφορά την ταχεία αντίδραση και την παρακολούθηση της αγοράς με απότερο σκοπό να βελτιωθούν οι ικανότητες ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση μελλοντικών κρουσμάτων. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ίσως περιθώριο βελτίωσης σε ό,τι αφορά την επικοινωνία από, από τις τοπικές τις κεντρικές αρχές, για παράδειγμα. Επίσης, ζητάμε μια επιστημονική μελέτη από την ΕΦΣΑ για την ε, αλυσίδα παραγωγής σε ό,τι αφορά α, την κατανάλωση σπόρων και Επιπλέον, Θέλουμε να εναρμονίσουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών από την βάση Β ε, σε ό,τι αφορά το μοριακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα διαφορά εργαστήρια μεταξύ της ΕΦΣΑ και του ECDC, του ΕΚΠΕΝ. Προφανώς ε, θέλουμε να γίνει και κάποια καλύτερη εκπίδευση σε ό,τι αφορά τα συστήματα αυτά και θέλουμε να συμμετάχουν και οι φορείς για την δημόσια υγεία και για την παρακολουθήση των τροφίμων. Αυτό ναι. αποτελεί σημαντική επιτυχή. Αυτά λοιπόν εν συντομία και φυσικά θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας σχόλια για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Μποκόνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση που μας δίνει πληροφορίες όσον αφορά την όλη προβληματική που δημιούργησε η ανησυχητική διάδοση αυτού του μικροβίου, του βακτηριδίου που πρέπει να μας απασχολήσει. Έχω κάποιες ερωτήσεις απλές. Πρώτη, μας λέτε κύριε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε να ζητήσουμε γνωμάτευση επιστημονική για να μειώσουμε τον κίνδυνο και τους κινδύνους σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, για αυτούς τους σπόρους που απαγορεύονται στην Ευρώπη. Για τα φύτρα του σιταριού. Λοιπόν, αυτά φορούν τη διατροφή. Υπάρχει στη διαδικασία της παραγωγής αυτών των βιολογικών σπόρων διαφορές σε σχέση με τη διαδικασία της παραγωγής ε, της συμβατικής που θα μπορούσε να εξηγήσει την ανάπτυξη του οίκολη. E. Με άλλα λόγια, τα βιολογικά προϊόντα λόγω της διαδικασίας παραγωγής είναι πιο επιρρεπή σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Κάναμε κάποιες μελέτες σχετικά με αυτό. Δεύτερον, είχαμε το Αμβούργο, Μπέγκλ στη Γαλλία και τη Λίλη. Βασικές πηγές μόλυνσης. Βασικές αιστείες όσον αφορά τη μόλυνση από τις φύτρες. Όσον αφορά τη Λίλ φαίνεται ότι ήταν ε, σε το είδος της παραγωγής ε, σε Χάμπουργκερ ότι ήταν η μόλυνση. Αυτή ήταν η πηγή της μόλυνσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα στην ανάλυση, να δούμε ε, το βακτήριο αυτό. Μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ακριβώς την πηγή και την πορεία αυτής της ε, μόλυνσης όσον αφορά τα τρόφιμα. Ευχαριστώ κύριο Κόνη, ο κύριος Σνέλχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ε, η παρουσίαση και έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας έχει ήδη εγκρίνει ψήφισμα όπου ε, αναφερθήκαμε στα προβλήματα και στα ερωτηματικά. Όλα αυτά καλά. Ένα συμπέρασμα μπορούμε να το βγάλουμε ήδη. Το όλο σύστημα έγκαιρης προεδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηθεί πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που ρώτησε η προλαλήσασα μας βασανίζει και μας έχουμε ξαφνικά πηγές μόλυνσης σε ένα τομέα που θεωρούσαμε ότι ήταν ασφαλέστατος. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βιολογική καλλιέργεια, στην οργανική, θα ορίσει πιο αυστηρούς ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι σημαντικό. In αλλά πιο σημαντικό είναι η κοινή γνώμη να γνωρίζει ε, κάπως περισσότερα για το πώς ε, παράγονται αυτά τα προϊόντα. 812 εκατομμύρια απώλειες. Γιατί όλος αυτός ο πανικός για τρόφιμα. Ε, αν εξηγούμε λίγο καλύτερα και με καλύτερη πειθαρχία και τάξη αν είχαμε δουλέψει, κυρίως οι πολιτικοί, γιατί οι ειδικοί, οι τεχνικοί, οι εμπειρογνώμονες ήταν πολύ καλοί, αλλά οι πολιτικοί από τις Βρυξέλλες να έχουμε περισσότερη επίρροη και στους πολιτικούς, να είμαστε λιγότερο λαϊκιστές γιατί πραγματικά θα πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη ε, και να είμαστε πιο ταχύ ε, στην αντίδρασή μας, να συνεργαζόμαστε με την επιστήμη. Κατά τα άλλα για την ομοθεσία, εντάξει, για τα μεταδοτικά νοσήματα. Α, θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσετε την εντολή να έχουμε εμβόλια πάντα διαθέσιμα, γιατί ε, ενώ ένα απόθεμα εμβολίων αυτό θα είναι πολύ ακριβό ή θα έχετε μια πάγια εντολή να δημιουργούνται, να παράγονται κάθε φορά ε, νέα εμβόλια. Γιατί είχαμε προβλέψει και ένα κονδύλι για εμβόλια για τη νέα γρήπη, τα οποία τελικά καταστράφηκαν, διότι δεν ε, απορροφήθηκαν. Σας ερωτώ στο μέλλον πώς θέλετε να το διχειριστείτε αυτό καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζανώνη. Και εγώ θέλω να τεθώ στο πρόβλημα το βιολογικό. Αυτό το γεγονός δημιούργησε κάποια σκιέα στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. Άκουσα καταναλωτές που ακόμα και τώρα βλέπουν να υπάρχουν ερωτηματικά και σκιές σε αυτό το τομέα. Πολύ επιβλαβή όλα αυτά για τον τομέα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός διότι συμβάλλει σε μια πιο καθαρή γεωργία που βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον με λιγότερα παρασιτοκτόνα και λιγότερα ε, λιπάσματα και άρα λιγότερες ε, εκπομπές που είναι επιβλαβές για το κλίμα. Υπάρχουν στοιχεία για όσον αφορά αυτή την αγορά για κάμψη σε αυτό το τομέα και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην μείνουν σκιές πάνω σε αυτό το τομέα αν έγιναν κάποιες σφιγμομετρήσεις όσον αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. όσον αφορά αυτό που συνέβη πριν από μερικούς μήνες και ποιες επιπτώσεις έχει όσον αφορά τον τομέα αυτών. Η κυρία Κόνη θέλει να προσθέσει κάτι, ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, σε αυτά που έλεγε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Νέλχαρτ, υπάρχει μια άλλη πτυχή όσον αφορά την κρίση που περάσαμε που συνδυάζεται με το e είναι η διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή διαπιστώσαμε ότι κάποιοι τομές δραστηριοτήτων υπέφεραν τα μάλα διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη και επειδή υπήρχε έλλειψη συντονισμού. Και διάφοροι κλάδοι, κυρίως της γεωργίας, ε, στις οικονομικές παρόλο που ίσως να μην επηρεαζόταν άμεσα από τη διάδοση αυτού του βακτηρίου. Θα πρέπει και αυτό να το εξετάζουμε την ασφάλεια τροφίμων και τη δημόσια υγεία, την προστασία του καταναλωτού, αλλά λάβουμε υπόψη και να προβλέπουμε πώς μπορούμε να χειριζόμαστε διαφορετικά τις κρίσεις για να υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες εκείνες που απαιτούν κάτι τέτοιο, που χρειάζονται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, θα σας δώσω το λόγο. Και θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε συγκεκριμένα στις δύο ερωτήσεις της κυρίας Οκονή, που είναι διαφορετικές. Από τη μια, ακριβώς πώς να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης ή της πρόληψης, λέει ο κύριος Σνέλχαρτ, ότι χρειάζονται επιστημονικές μελέτες, αλλά όταν η κατάσταση είναι πήγουσα, τι κάνουμε και η δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με αυτό είναι η διαχείριση της κρίσης. Να προσπαθήσουμε να έχουμε μια διαχείριση ίσως πιο ισόρροπη που να λαμβάνει υπόψη και τα γεωργικά συμφέροντα αλλά και την ανασφάλεια στην οποία βρισκόμαστε τη στιγμή που ξεσπάει αυτό το κρούσμα και έχουμε και θύματα και απώλειες διαδοχικές ανθρωπίνων ζώων. Είναι περίπλοκα αυτά τα θέματα και τα ξέρουμε. Αν μπορούσατε να μας διαφωτίσετε λίγο περισσότερο γι' αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε στα μέσα της ε, ε, αξιολόγησης και όπως ανακοινώσαμε τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε εφόσον θα έχουμε ε, την απαραίτητη επιπρόσθετη ενημέρωση και από την ΕΦΣΑ αλλά και από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και τις εμπειρίες τους. Δηλαδή, τι σας λέγω τώρα. Αυτά που σας αναφέρουμε τώρα δεν είναι οριστικά, δεν είναι τα τελικά στοιχεία, διότι είμαστε ακόμα στη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων και διδαγμάτων. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στο εξής. Είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε σε όλους ότι ε, τα κρούσματια κόλλη κανονικά ε, γαστρεντερίτιδες ε, εμφανίζονται στην Ευρώπη ε, κάθε χρόνο και κατά χιλιάδες. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ειδικό στέλεχο, μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση. Οι γαστρεντερίτιδες που οφείλονται στην εσερίχια κόλλη είναι αρκετά συχνέ κατά τα άλλα. Και πρέπει να σα πω ότι ε, η υπόθεση της Λίλης ήταν διαφορετικό στέλεχος και δεν είχε καμία επαφή με την άλλη υπόθεση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να συνδέουμε αυτά τα δύο γεγονότα και τις δύο περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βιολογική παραγωγή, την οργανική γεωργία. Αν είναι αρκετά ασφαλή ή όχι και τι πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να πω και πάλι ότι συνεχίζει η ανάλυση, αλλά οφείλω να πω το εξής. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα ε, στους σπόρους ε, τριγωνέλα από mm. την Αίγυπτο, θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι σπόροι δεν προορίζονταν ε, αρχικά ενδεχομένω για ανθρώπινη κατανάλωση και από τέτοιου πόρους παρήχθησαν φύτρα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ το ζήτημα αν είναι βιολογική γεωργία ή άλλη, αλλά να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Θα πρέπει να ελέγχονται τα πάντα και αυτέ οι περιπτώσει κάποιοι σπόροι που φυτρώνουν και τα φύτρα μπαίνουν στη τροφική αλυσίδα της ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό θα πρέπει να ελέγχονται. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη κρίση, βεβαίω και συμφωνώ με όλου σα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό στοιχείο. Και πάλι όμω χωρί σωστή ανάλυση είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανεί ε, για το ποια είναι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης. Όπως σας είπα, καμιά φορά κυκλοφόρησαν πληροφορίε που δεν ήταν τελείως τεκμηριωμένες ή στοιχειοθετημένε επιστημονικά. Αυτό οδήγησε στην υπερβολική καμιά φορά αντίδραση του κοινού, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε και να αναλύσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι, προφανώς. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχίζει κάποια συγκεκριμένη δεδομένη χρονική στιγμή. Και εμεί θα πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σα θυμίσω μόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν... Uh, θα πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο τις πληροφορίες για να είμαστε σε θέση να πούμε ποια ακριβώς διδάγματα μπορούμε να εξάγουμε από τη συγκεκριμένη περίπτωση. <clears throat> Θα παρακαλέσω ακόμα τον συνάδελφό μου να σας δώσει Ορισμένε απαντήσει στις ερωτήσει σα για τη δημόσια υγεία. Από πλευρά δημόσια υγεία και όσον αφορά τη διαχείριση των ε, κινδύνων, να πω ότι αυτό το γεγονό με το E. έδειξε ότι ήταν η πρώτη φορά που οι εκείνοι που διαχειρίζονται κίνδυνο, το δημόσιο κίνδυνο όσον αφορά την υγεία συναντήστηκαν με συναδέλφους τους και βάσει των διαφόρων εντολών των αρμοδίων επιτροπών Ταυτόχρονα υπήρχαν ε, διασκέψεις, τηλεδιασκέψεις καθημερινά για να βλέπουν πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα από πλευράς δημόσιας υγείας, κοιτάζοντας τα στατιστικά στοιχεία, τις πρόσφατες πληροφορίες που κατέφθαναν από πλευράς δημόσιας υγείας και δεύτερον εξετάζοντας τι μέτρα θα μπορούσαν να ε, εφαρμοστούν από πλευράς δημόσιας ε, προστασίας υγείας από άτομα τα οποία είχαν ε, προβλήματα με τα νεφρά του χάρη και να εντοπίζουμε πλευράς ερωτηματολογίων ε, προς τους ασθενείς την πηγή του προβλήματος για όσοι είχαν πρόβλημα ανεπάρκεια νεφρών και από πλευράς των διαφόρων ε, εκοσώπων του ιατρικού τομέα να γίνει μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ νοσοκομείων και γιατρών που ε, θεράπευαν τους ασθενείς. Όλα αυτά γινόταν σε πραγματικό χρόνο. Κάθε φορά, σε κάθε συνεδρίαση υπήρχε και παρέμβαση συναδέλφων της Υπηρεσίας Ασφαλείας Τροφίμων και βλέπαμε πληροφορίες που συνέλεγαν αυτής από τα εργαστήρια από την πλευρά της ασφαλείας τροφίμων και προσπαθούσαν να δουν τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αποσυρθούν προϊόντα από την αγορά. Ήταν ενδιαφέρον το πείραμα αν θέλετε όσον αφορά τη συνδιαχείριση μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτικών. Δημόσια υγεία με την πλευρά με πολύ περιορισμένες νομικές εξουσίες και τη πλευράς ασφάλεια τροφίμων με πολύ πιο ανεπτυγμένε ρυθμιστικέ και νομικές εξουσίες. Μετά όσον αφορά την επικοινωνία και τι ανακοινώσει, θα ήθελα να πω ότι από το 2009 από την πανδημία H1N1 θεώρησαν τα κράτη-μέλη ότι χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερο συντονισμό ε, ε, της με το κοινό και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου με το E. κινητοποίησαμε και την ε, Επιτροπή ε, Προστασίας της Υγείας, Ασφαλής της Υγείας για να εντοπίσει ποια μηνύματα κινούνται στο δημόσιο τομέα, ποια επικοινωνία υπήρχε μέσω των εφημερίδων ή μέσω του διαδικτύου με το κοινό και να προσπαθήσουμε να, να ετοιμαστούμε όσον αφορά την επικοινωνία για να δίνουν πληροφορίες βάσει της ε, πιο πρόσφατης επιστημονικής εικόνας. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επισημοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας, όπως είπα και στην αρχή, και αυτό σαν πλαίσιο της πρωτοβουλίας ε, για την ασφάλεια της υγείας που εξετάζαμε φέτος. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι βασική πτυχή η επικοινωνία της διαχειρίσεως του, του κινδύνου και θέλουμε αυτό να το επισημοποιήσουμε και να επισημοποιήσουμε αυτή τη δομή αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σνέλχαρτ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ναι, θα ήθελα να θέσω μια επιπλέον ερώτηση. Ίσως κάτι να κατάλαβα λάθος, αλλά είπατε ότι τα φύτρα που είχαν εισαχθεί δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα. Όχι. Παράγουμε όμως ένα προϊόν το οποίο καταλήγει στα τρόφιμα και είπατε ότι δεν υπήρχε σχετική έγκριση, μα πρόκειται για ποινικό αδίκημα στην περίπτωση αυτή. Για ποιο σκοπό έγινε η εισαγωγή λοιπόν του σπόρου. Ο σπόρος ο οποίος δεν περιλαμβάνει. Γιατί απαγορεύτηκε για την παραγωγή τροφίμων αυτός ο σπόρος. Αυτό δεν το κατάλαβα. Θα θέλετε να το διευκρινίσετε παρακαλώ. Θα μπορούσε ένας από τους δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ναι. Καλησπέρα σας. Όχι, οι σπόροι αυτοί, το πακέτο ήταν για σπορά και όχι, δεν προοριζόταν για ανθρώπινη κατανάλωση. ο σκοπός ήταν να χρησιμοποιηθούν τα φύτρα τα οποία θα προέκυπταν στο κρούσμα στη Γαλλία. Εντοπίστηκε η προέλευση από ένα συγκεκριμένο τέτοιο πακέτο για σπορά. Bon, bah écoutez, euh, Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, κυρία Κόνη, εγώ είμαι καταναλώτρια αυτών των προϊόντων. Είναι μικρά φυτόργια, πουλώνουν μικρές συσκευές για την κουζίνα που πολλούνται. Με τα προϊόντα που θα μπορούν να φυτρώσουν και με και να μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί σαν φύτρα για διακόσμηση πολύ συχνά. Και από τη στιγμή που έχουμε καταναλώσει ε, τους σπόρους που είναι σε αυτό το μηχανισμό ε, για να φυτρώσουν, αγοράζουμε εκτός τη συνολική αγοράς των σπόρων. λένε αυτέ οι σπόροι ότι είναι μόνο για φύτεμα και όχι για κατανάλωση. Οπότε αυτό πώς μπορεί να διαπιστωθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν λένε ποτέ ότι δεν πρέπει να καταναλωθούν αυτοί οι σπόροι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά και εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στι 27 Οκτωβρίου στι 9 η ώρα στο Στρασβούργο. Σα εύχομαι μια έξοχη βραδιά. Καλό σα βράδυ.